Liebe Kolleginnen und Kollegen, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω ενθέρμως τον υποψήφιο υπο... Επίτροπο για τα θέματα μεταφορών, τον κύριο Μάρο Σέσκοβιτς. Και θέλω να σας ότι ο στόχος της σημερινής ε, ακρόασης βάσει του κανονισμού μας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να κρίνει τον ε, υποψήφιο από τη βάση της ικανότητάς του, της δέσμευσή του σε σχέση με την ευρωπαϊκή ιδέα και της ανεξαρτησίας του. Φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και τις γνώσεις του στον τομέα του επιστητού που θα αναλάβει και την ικανότητα επικοινωνίας του. Θέλω περαιτέρω να αναφέρω ότι στην, ε, στην ακρόασή μας θα λάβουν μέρος και βουλευτές από την Επιτροπή Ήτρα για να θέσουν ερωτήματα σε σχέση με τη διαστημική πολιτική. Η Ήτρε λοιπόν συμμετέχει σε αυτή την ακρόαση. Επίσης θέλω να σας πεθυμίσω ότι ο κύριος Εύκοβιτς έχει δώσει γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε και οι ερωτήσεις αυτές και καθώς και απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στους βουλευτές. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Πρωτού λοιπόν δώσω το λόγο στον υποψήφιο κύριο Επίτροπο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να κάνω κάποιες διαδικαστικού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Η ακρόασή μας θα ακολουθήσει την μέθοδο ping-pong. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ερώτηση θα ακολουθηθεί από μία απάντηση. Θα έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο πρώτος αφορά τους συντονιστές, με συνολικό χρόνο 5 λεπτά για κάθε ερώτηση. Για όλους τους άλλους βουλευτές ο χρόνος θα είναι 3 λεπτά. Και να λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ στενός. Επομένως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι θα εμφανίζεται ο χρόνος, η αντίστοφη μέτρηση στις οθόνες. Εγώ θα διακόψω όποιον ξεπερνάει το χρόνο του και αυτό ισχύει και για τον υποψήφιο κύριο Επίτροπο. Παρακαλώ να τηρήσετε λοιπόν το χρόνο ομιλία σας. Στον πρώτο γύρο θα έχουν οι συντονιστές 5 λεπτά σύνολο. Μπορούν να θέσουν μια ερώτηση το πολύ 2 λεπτών και ο αρμόδιος, ο υποψήφιος επίτροπος θα πρέπει να απαντήσει. Έχει χρόνο να απαντήσει τρία λεπτά το maximum. Να έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας, ότι όσο μακρότερη είναι η ερώτησή σας, τόσο πιο σύντομη θα είναι η απάντηση του Επιτρόπου. Εν τη συντομία η αρετή. Εάν λοιπόν δεν, υπάρχει, δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος των πέντε λεπτών, θα υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής ερώτησης. Αλλά οι συμπληρωματικέ ερωτήσει δεν μπορούν να διεξέλθουν άλλο θέμα από αυτό τη αρχική ερώτηση. Δεν μπορούν να εισαγάγουν ένα νέο θέμα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ ω πρόεδρο θα είμαι υποχρεωμένο να διακόψω και να αναλάβω να αφαιρέσω το λόγο από τον αρμόδιο συντονιστή. Στο δεύτερο γύρο θα έχουν οι βουλευτές τρία λεπτά για ερώτηση και απάντηση. Και εδώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο σύντομη είναι η διατύπωση ερώτησης, τόσο περισσότερο χρόνο έχει αρμόδιος ο Επίτροπος για να δώσει μια πλήρη απάντηση. Στον δεύτερο γύρο μπορεί να επιτραπεί μια συμπληρωματική ερώτηση εάν παραμένει τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την πρώτη ερώτηση και απάντηση. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ο κάθε ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν τη δική τους γλώσσα και φυσικά και ο υποψήφιος κύριος Επίτροπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει διερμηνία, μην μιλάτε πολύ γρήγορα, ώστε να έχετε πλήρη διερμηνία των λόγων σας. Η συνολική ε, ακρόαση βρίσκεται στο διαδίκτυο στην, ε, σε web streaming και θα εμφανιστεί αργότερα και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και στο Twitter, στο hashtag EPHearings2014 μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τεκτενόμενα. Και τώρα μετά από αυτές τις διευκρινήσεις θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαροσεύκοβιτς, τον υποψήφιο επίτροπο, για 15 λεπτά το maximum να κάνει τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις προς την Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας κύριε ε, Σεύκοβιτς και για τις δηλώσεις σας για το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη, ώστε να υπάρξει πραγματικά προστασία της κινητικότητας αλλά και του κλίματος. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Κύριε Πρόεδρε, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, μου εξηγήσατε πόσο σημαντικό είναι για σας το να υπάρχει ένα αηφόρο σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Και μου μιλήσατε για την στράτευσή σας για ένα ευρωπαϊκό ποδηλατόδρομο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχουμε εργαστεί και οι δύο έχουμε ζήσει και οι δύο από τις δύο πλευρές του σιδηρού παραπετάσματος, εγώ στην Πρατισλάβα, μια εποχή όπου δεν μπορούσε ε, κανένας νέος να φανταστεί το μέλλον του μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, έχουμε ζήσει μια ιστορική μετάλλαξη τα τελευταία 25 χρόνια και ιδιαίτερα από τον ψυχρό πόλεμο και την, ε, το διχασμό της Ευρώπης είχε πληγεί ο τομέας των μεταφορών και γι' αυτό προτεραιότητά μου θα είναι να ε, αντιμετωπίσω τις διαφορές, τα προβλήματα, τις ασυμβατότητες στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι όπως και εσείς, ε, ήμουν υποψήφιο και εγώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξελέγην βουλευτή. Είχα και εγώ, όπω και εσεί, την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλού πολίτε σε αυτή τη διαδικασία και έτσι γνωρίζω πολύ καλά ποιοι είναι οι τομεί τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που του ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Οι πολίτε λοιπόν σε αυτέ τι συνομιλίε επιβεβαίωσαν ότι οι μεταφορέ ένα καλό δίκτυο υποδομών των μεταφορών, ένα καλώς λειτουργούν σύστημα των μεταφορών, ε, είναι απαραίτητο και έχει την ευθύνη για την ε, ανάπτυξη των διευρωπαϊκών διαδρόμων των μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αποδείξουμε ότι πρόκειται για μια από τις καλύτερες αποδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στις μεταφορές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι μεταφορές και η κινητικότητα είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη στον 21ο αιώνα αξίζει ένα σύστημα υψίστου επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου των μεταφορών, εάν θέλουμε να παραμείνουμε ηγετικοί, ε, ε, στην ηγετική θέση ανά τον κόσμο θα πρέπει να έχουμε και περιβαλλοντικά και οικολογικά σωστές μεταφορές αλλά και ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές και επιμελητία Έτσι λοιπόν η οικονομική, και καθώς η οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία αξιοπρεπών και ε, αηφόρων θέσεων εργασίας είναι προτεραιότητα υπαριθμών ένα για την Επιτροπή της του... του Πρόεδρου Γιούνκερ, πιστεύω ότι οι κοινέ μας προσπάθειες στον χώρο των μεταφορών ε, και το διάστημα μπορούν σημαντικά να συμβάλλουν στο στόχο αυτό. Ε, περιμένω λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε ώστε να αναπτύξουμε το πακέτο των ε, επενδύσεων για 300 δισεκατομμύρια ευρώ με μια καινοτόμο προσέγγιση που θα σημάνει μόχλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών υποδομών με καλά σχέδια, με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να βγάλουμε την Ευρώπη, έξω, να την βγάλουμε την Ευρώπη από την κρίση και να τη φέρουμε πιο κοντά σε ύψη του επίπεδου υποδομέ για τον 21ο αιώνα όπω τι χρειάζεται και πρέπει αυτό να το κάνουμε ένα σαφέ όραμα. Πρέπει να ετοιμάσουμε την Ευρώπη όχι για αυτό που χρειάζεται σήμερα, αλλά για αυτό που θα έρθει στο μέλλον, δηλαδή για αυτό που θα χρειαζόμαστε σε 10, 20 και 30 χρόνια στι μεταφορέ. Άρα χρειάζεται να αναπτύξουμε φυή συστήματα μεταφορών, χρειάζεται να εργαστούμε σε πλήρω ε, διατροπικά, ολοκληρωμένα δίκτυα, στηριζόμενα στι νέε τεχνολογίε, τι δορυφορικέ και τι ψηφιακέ. Χρειαζόμαστε νέε υπηρεσίε και προϊόντα, τα οποία θα επιτρέψουν στου Ευρωπαίου πολίτε και τι επιχειρήσει να έχουν την επιλογή αηφόρων μεταφορών, ε, τρόπων μεταφορών που θα μπορούν με ένα απλό πάτημα του κουμπιού σε ένα FES τηλέφωνο να ε, χρησιμοποιούν. 70% των ε, πολιτών λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν ε, σε αστικά κέντρα και ως εκ τούτου οι μεταφορές όλο και περισσότερο επηρεάζουν τη ζωή, τη ζωή τους είτε πρόκειται για την επιλογή του βαδίσματος, του ποδηλάτου, της οδήγησης ενός αυτοκινήτου ή της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα μεταφορών στηριζόμενο στις πιο καινοτόμε λύσεις που θα δώσει και στην Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της πάλι, που θα εξασφαλίσει ε, θέσεις εργασίας, αυτό που ονομάζουμε cool jobs, ωραίες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους και θα εξασφαλίσει σταθερότητα για, το ένα, ε, για τα 11 εκατομμύρια των εργαζομένων στο χώρο των μεταφορών που αυθουσιώνουν τη ζωή τους σε αυτό. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ασφάλεια και την, ε, τις συνθήκες αποφυγής κινδύνων. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το όραμα στο οποίο αναφέρομαι. Αναφέρθηκα στο δίκτυο των TNT το δίκτυο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών δηλαδή, τα οποία θα πρέπει με ιδιαίτερη έμφαση να, να εφαρμόσουμε, με ιδιαίτερη αυστηρότητα, να χρησιμοποιήσουμε ε, όλους τους διαδρόμους και σκοπεύω να ξεκινήσω με τις νομοθετικές προτάσεις που ήδη βρίσκονται επιτάπητος, όπως το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους, τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, ε, μέτρα δηλαδή και ρυθμίσεις τα οποία πιστεύω μπορούμε να εξασφαλίσουμε σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχω πλήρη επίγνωση των κοινωνικών ευαισθησιών των ε, ανησυχιών σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η πρότασή μου για να τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα ζητήματα θα ήταν να εμπαθύνουμε στον ε, κοινωνικό διάλογο, να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δούμε πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία των μεταφορών, αλλά όχι ει βάρο των ε, εδρεωμένων κοινωνικών προτύπων και προδιαγραφών. Οι περισσότερε από τις θετικέ εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μεταφορές Ευρωπαϊκής Ένωση δεν είχαν εξασφαλιστεί εάν δεν υπήρχε και ύψιστο επίπεδο ε, δικαιωμάτων των μεταφορών για κάθε είδο μεταφορών. Είμαι βέβαιο ότι αυτό αποτελεί και το κλειδί ε, ώστε να εξασφαλίσουμε όπως καταφέραμε τελικά να σταματήσουν οι πρακτικές των εταιριών που είχαν να κάνουν με το overbooking ή τις αλλαγές προγράμματος και διαδρομών της τελευταίας στιγμής. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ο ενιαίος χώρος των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε τρόπο μεταφορών και τους σιδηροδρόμους ασφαλώς με την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων όπως το RTMS για τη, ε, ε, συστημάτων σήματος που υπάρχουν ήδη σαν δυνατότητες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων ώστε να απαλλαγούμε από τις 26.000 διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα αυτού και, την χρήση, και να προχωρήσουμε στην χρήση κοινών ε, επιχειρήσεων ε, όπως το Shift to Rail για να σχεδιάσουμε διατροπικούς ε, σιδηροδρόμους για το μέλλον. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε έτσι αξιόπιστη παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, ύψης της ποιότητας και ε, οικονομικές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα βοηθήσουμε και τους, τον κατασκευαστικό κλάδο των υποδομών των σιδηροδρόμων. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι πιστεύω ακράδαντα το όρο του ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων. Δεν μπορούμε να χάνουμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο επειδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο και ως εκ τούτου να πιέζουμε τα αεροπλάνα μας να παίρνουν πιο μακρινά δρομολόγια που κοστίζουν και περισσότερα αλλά και παράγουν περισσότερα, εκπέμπουν περισσότερα ε, αέρια ε, του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να εργαστούμε και για την αποδοτικότητα των αδρομίων μας και για τη δυνατότητα να κοιτάξουμε, να στραφούμε προς την ε, γειτονία μας όπως η παραδείγμα τη Μέση Ανατολή όπου υπάρχει σημαντική, σημαντικός ανταγωνισμός. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να μην χάσουμε την, το δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πολύ μεγάλη δουλειά μπορεί να γίνει από το ΣΕΤΑΡ και τις του που πιστεύω μαζί με το δυναμικό που έχουμε σε δορυφορική συστήματα μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας ε, και του εξεχρονισμού αυτού του κλάδου. Όπως γνωρίζετε η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός, ε, το μεγαλύτερο εμπορικό σύνολο στον κόσμο. Όλες δεν γνωρίζουμε, δεν θυμόμαστε μερικές φορές το 75% των μεταφορών μας ε, είτε πρόκειται για εξαγωγές είτε πρόκειται για εισαγωγές περνάνε από τα πλοία. 40% των παγκοσμίων των πλοίων όλου του κόσμου ανήκουν σε ευρωπαϊκά χέρια, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι η μεγαλύτερη μεγαλύτερη ε, διάβλη ε, θαλασσίων μεταφορών στον πλανήτη. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο και στον τομέα αυτών. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το τομέα αυτό, όπω και άλλοι, θα εξασφαλίσει πλήρη ολοκλήρωση και διατροπικότητα μέσα σε έναν νέο ευρωπαϊκό χώρο των μεταφορών. Αυτό σημαίνει εξυγχρονισμό των υποδομών των ε, λιμένων και ένα σύστημα μεταφορών χωρί φραγμού. Πρέπει να βρούμε επίση αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη ατμοσφαιρική ρήπανση, γιατί όπου μιλάμε για ένα παγκόσμιο κλάδο οικονομία, οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουμε και στο πλαίσιο τη Παγκόσμια ναυτιλιακής Οργάνωση και αντίστοιχα για τι αεροπορικέ μεταφορέ, τη ΙΚΑΟ, ε, των οποίων είναι και μέλη τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία λοιπόν μας από τα κέντρα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση επίση στου ιστορικού πλωτού δρόμου που πολύ συχνά μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη λύση σχέση με τα προβλήματα της ρήπανσης, της, ε, του δυναμικού και της προσβασιμότητας. Αλλά αυτός ο κλάδος ε, είναι κατακαιρματισμένος με στόλο απαρχαιωμένο και πολλές φορές ε, πλωτές οδούς που δεν αξιοποιούνται, όπως ο Δούναβης που είναι μόνο στο 15% του δυναμικού του. Με το πρόγραμμα Ναϊάδες τώρα μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή σε αυτόν τον κλάδο και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν καλύτερα και να εργαστούν πιο ανταγωνιστικά στον χώρο αυτό. Αν μου επιτρέπετε κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το tour de monde όπω το λέμε, αυτή την επισκόπηση με τις οδικές μεταφορές. 72% των ε, μεταφορών γίνονται με αυτοκίνητο, 40% των φορτίων ε, μεταφέρονται με φορτηγά, τεράστιος κλάδος λοιπόν και με σημαντικές προκλήσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως καλύτερη οργάνωση των οδικών μεταφορών ώστε να μην συνεχίσουμε το φαινόμενο να ταξιδεύουν ένα στα τέσσερα φορτηγά μας άδεια στους δρόμους μας ενώ ταυτόχρονα χάνουμε 1% του ΑΕΠ μας ε, λόγω της συμφόρησης. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και ως προς την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει για να διατηρήσουμε την, ε, τις υποδομές μας σε καλό επίπεδο και να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τις εργασίες μας επίσης να κοιτάξουμε ε, να αναζητήσουμε έναν πιο εμβαθισμένο και συνολικό τρόπο για τις διαφορετικές εφαρμογές του συμφωνημένους ε, τρόπους όπως είναι κανόνες όπως είναι η αρχή του Καμποτά. Η πίεση προς τον κλάδο για τον περιορισμό των συμφορήσεων της, ε, ε συγχωρήπανσης και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει και την ασφάλεια. Είμαι αποφασισμένος ότι θα, θα αγωνιστώ για το θέμα αυτό γιατί πιστεύω ότι κάθε πρόοδο στον τομέα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον αριθμό των ε, δυστυχημάτων, των τροχιών δυστυχημάτων κάθε χρόνο. Με 26.000 ε, δυστυχήματα το χρόνο έχουμε υπερβολικά υψηλά ποσοστά. Πιστεύω ανα, ε, απαράδεκτο αυτό και για μένα και για σας. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα για συμβασμό προς το θέμα της ασφάλειας σε κάθε τρόπο μεταφορών και η Ευρώπη θα καταστεί ο πιο ασφαλής χώρος μεταφορών στον κόσμο. Είμαι πεπισμένος ότι πολύ γρήγορα θα δούμε και περισσότερα ευφυή οχήματα στους δρόμους μα που θα μπορούν να επικοινωνούν, να μιλάνε το ένα με το άλλο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικέ μορφές ενέργειας ε, με, ευρωπαϊκού, ε, με ευρωπαϊκές εμβέλειες υποδομές. Αυτό σημαίνει βεβαίως το μέλλον για τον, οδικό, για τον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά για να επιτύχουμε του στόχου αυτού, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα κανονιστικό πλαίσιο και ευρωπαϊκέ υποδομέ Για το, και για το... Χαίρομαι λοιπόν. Βλέπω ότι συνδέονται εκ νέου το διάστημα και οι μεταφορές. Το διάστημα έρχεται πιο κοντά στους χρήστες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα επόμενα έτη θα είναι κρίσιμα για τη διαστημική Ευρώπη. Μέχρι το 2020 ο στόχος μας είναι να έχουμε τις υπεύθυνε υποδομές στο διάστημα για να δώσουμε υπηρεσίες μέσω του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικους. Για να το πετύχουμε θα θέσουμε σε κυκλοφορία πάνω των 30 δορυφόρων τα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ιδιαίτερα προχωρημένη τεχνολογικά. Τα διαστημικά προγράμματα της Ένωσης θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της, θα δώσουν κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία και θα δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης υψηλού επίπεδου. Να μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως το διάστημα είναι στην υπηρεσία των πολιτών όταν χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, όταν κάνουν συναλλαγές οικονομικές, όταν παίρνουν το αεροπλάνο, όταν βλέπουν ειδήσει για τον καιρό ή ψάχνουν το πιο κοντινό ε, εστιατόριο μέσα από το αυτοκίνητό τους, χρησιμοποιούν τις διαστημικές υποδομές. Το 7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εξαρτάται από τις διεθνείς εφαρμογές ε, κυκλοφορίας ε, και ρύθμισης από πλευράς των δορυφόρων. Βέβαια όλα αυτά είναι δύσκολα να τα πετύχουμε, ε, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Το ατύχημα το οποίο συνέβη ε, στα πλαίσια του δορυφόρου για τον Καλλιλέο τον Αύγουστο δεν πρέπει να μας απογοητεύει, αντίθετα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό και να του δώσουμε μια νέα όθηση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, οι μεταφορές είναι ένας τομέας ο οποίος φύγει τους πάντες, αφορά καλύτερα τους πάντες. Είναι ο σκελετός αν θέλετε της σύγχρονης κοινωνίας. Οι επιμελητιακές λειτουργίες και οι μεταφορές γενικά στηρίζουν κάθε μορφή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Εφόσον με επιβεβαιώσετε θα συνεργαστώ μαζί σας έτσι ώστε να, να ενισχύσουμε αυτήν την ηγετική θέση της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα, να δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, καινοτομία να προχωρήσουμε και να φυσικά προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε σας ευχαριστώ γιατί δείξατε και τις γλωσσικές σας ικανότητες χρησιμοποιώντας πολλές γλώσσες και χαίρομαι και για το γεγονό ότι χρησιμοποιήσατε και τη μητρική μου γλώσσα τα γερμανικά. Έρχομαι τώρα στους συντονιστές. Ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν μιλάτε ακόμα Ολλανδικά, αλλά νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚ. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας με ένα φιλόδοξο και δίκαιο τρόπο. Χωρίς τις μεταφορές όλα είναι στατικά. Φυσικά ακόμα και η, η ευρωπαϊκή ιδέα. Έχω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, η λευκή βίβλος για τον οδικό χάρτη για μια ενιαία ζώνη μεταφορών στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ορισμένε προτεραιότητε, τι οποίε τι αποδέχεστε εσεί ή όχι. Θέλετε να τι αλλάξετε, ποια είναι τα σχέδιά σα για το θέμα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Η χρηματοδότηση των σχεδίων TEN-T. το αναφέρατε αυτό. Μιλάτε για 300 δισεκατομμύρια από τον κύριο Γιούνκερ που έχουν αναγγέλθει Πόσα από αυτά τα 300 δισεκατομμύρια όμως θα αφιερωθούν στα προγράμματα και τα σχέδια του ΤΕΝΤΗ. Θα θέλαμε να έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Και τέλος ένα πιο δύσκολο σημείο. Η συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους και τους άλλους γενικούς διευθυντές. Έχουμε σημειώσει ότι ο Επίτροπος Μεταφορών βρίσκεται πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τον Επίτροπο Ανταγωνισμού, τον Επίτροπο ε, <clears throat> Περιβάλλοντος κτλ. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα, γιατί οι μεταφορές πρέπει να παίξουν ένα προεξέρχοντα ε, ρόλο στην κοινωνία μας. Και τέλος, επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, θα ήθελα να σας, πω, να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για αυτούς που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Μιλήσαμε για αεροπλάνα, για τρένα, για μεγάλα σχέδια. Τι θα κάνετε όμως για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Θα κλείσω εδώ, δεν ήθελα να ε, πάω πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Θα βελτιώσω τα Ολλανδικά μου, σας το υπόσχομαι. Για να έρθω στα ερωτήματά σας. Όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τον οδικό χάρτη για τα επόμενα πέντε χρόνια, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ότι όσο πιο σύντομα έρθει η μεταρρύθμιση της Λευκής Βίβλου, τόσο και καλύτερα. Γιατί πιστεύω ότι το δίδαγμα των τελευταίων ετών ήταν ότι ήταν κάπως καθυστερημένα η Λευκή Βίβλος στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά έπρεπε να τροποποιηθούν τα σχέδια για νομοθεσία. Σας υπόσχομαι λοιπόν θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να επιταχύνω τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Λευκής Βίβλου. Μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι η πρόοδος για το σχέδιο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική. 24 από 40 δράσεις που προβλεπόταν στη Λευκή Βίβλο έχουν ήδη ή περατωθεί ή ξεκινήσει. Και φυσικά είμαι έτοιμος να τα συζητήσω και με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν, γιατί αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί από το σύνολο της Επιτροπής και μετά θα επανέλθει σε εσά και θα σας ζητήσει η Κομισιόν να το επεξεργαστείτε μαζί μας. Για τα σχέδια TNT και τα 300 δισεκατομμύρια, τις επενδύσεις των 300 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ότι 26 δισεκατομμύρια για τα σχέδια TNT είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι μια σταγόνα εν το ωκεανό. Αν δείτε τι χρειάζεται η Ευρώπη, χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι καλά σχέδια υποδομών, σχέδια που ευνοούν την μελλοντική ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων είναι σχέδια όπου μπορούν να υπάρχουν και πολλές προοπτικές για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Μπορούμε λοιπόν να προωτήσουμε αυτή την εταιρική σχέση δημόσιου ιδιωτικού τομέα και να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει επιτευχθεί και χάρη στη δική σας συμβολή μέσα στις ε, νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ακριβώς πώς θα γίνει αυτό και πόσο ποσοστό αυτό των κονδυλίων θα πάνε στη δημιουργία υποδομών είναι δύσκολο να σας το πω τώρα, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε εξίσου ελκυστικά σχέδια για εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που ε, επιτυγχάνει αυτή η εταιρική σχέση. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία με όλους τους ε, συναδέλφους στην Κομισιόν και τους αντιπρόεδρους και οι ανάδρομες ροές ε, και αυτές είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Τίσεν θα δώσει μια απάντηση πιστεύω για τα θέματα προσβασιμότητας που περιλαμβάνει και τα προβλήματα των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Σας ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου και περνάμε στον επόμενο ομιλητή, ονόματο της Σοσιαλιστικής Ομάδο τον κύριο Έρτουχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάθε επιτυχία από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Έρχομαι στο πρώτο μου ερώτημα τώρα που έχει να κάνει με το κοινωνικό δίκαιο και τα θέματα της εφαρμογής του. Τις κοινωνικές πτυχές τις θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα να ξέρω αν συμφωνείτε ότι η διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωση και αν συμφωνείτε αν θέλετε πράγματι να τα εφαρμόσετε και στην πράξη. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα της λεγόμενης βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Βλέπουμε ότι στις πόλεις υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση για τις μεταφορές και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πώς ε, ε τοποθετήστε σε σχέση με την ε, τωρινή πολιτική κινητικότητα της πόλης που βλέπετε σφάλματα και που θεωρείτε πρέπει να υπάρξουν τροποποίησεις ο διαμεσ... η, το... Ε, η από κοινού χρήση αυτοκίνητο παραδείγματος χάρη είναι ένας σημαντικός ε, χώρος. Ε, μπορεί η Κομισιόν να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα αυτό και στην δημόσια, δημόσιες μεταφορές και όχι μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τις λιμενικές, τα λιμενικά θέματα. Το πακέτο για την πρόσβαση στα λιμάνια και την ε, διαφάνεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό και αυτό συνάπτεται με τις κρατικές επιδοτήσεις. Πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς τις προσπάθειες για να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τις υποστηρίξεις και πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα αναχαιτιστούν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και έρχομαι τώρα στα λεγόμενα μεγάλα ε, για τα ε, μεγάλα πλοία και επίσης αν θα μπορέσει η Κομισιόν να προωθήσει νέα νομοθεσία για, την, ε, για το συνδρομικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Θα προσπαθήσω να απαντήσω τηλεγραφικά γιατί θέσατε πάρα πολλά θέματα ταυτόχρονα. Καταρχάς σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πράγμα ισχύει. Όταν προετοιμάζουμε τις νομοθετικές προτάσεις και όταν τις βάζουμε σε αξιολόγηση για την μελέτη των επιπτώσεων το ερώτημα το οποίο πρώτα θα τίθεται είναι το πώς αυτό θα επηρεάσει την απασχόληση στην Ευρώπη. Θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης ή θα δημιουργούμε προβλήματα ε, στους εργαζομένους. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αρχή την οποία πρέπει να σεβαστούμε και στον τομέα των μεταφορών. Για να είμαι ειλικρινής και βλέποντας το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε καλύτερα σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο. Γνωρίζω ότι διεξάγεται ο κοινωνικός διάλογος. Γνωρίζω ότι κυρίως οι συζητήσεις γίνονται σε τεχνικό επίπεδο και για να δημιουργηθεί ε, αν θέλετε περισσότερο, ένα καλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης απαιτείται περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Τώρα, για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες γενικά. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε αφήσει πίσω μας δύσκολες στιγμές. Υπάρχει τώρα πλέον μια τρίτη πρόταση για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Θα συνεργαστώ μαζί σας και με τους κοινωνικούς εταίρους για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των λιμένων. Γιατί είναι πραγματικά οι θύρες της Ευρώπης και απαιτείται να τις συνδέσουμε με τα Τέν, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όχι μόνο σε σχέση με τους τρεις λιμένες ε, ε, στους οποίους αναφέρθηκα ήδη, αλλά το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων. Τώρα, για την αηφορία στις αστικές μετακινήσεις. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ζουν στις πόλεις και τα περισσότερα ατυχήματα ε, γίνονται στην πόλη, οι εκπομπές είναι περισσότερες στις πόλεις. <clears throat> Είναι λογικό λοιπόν να υπάρξουν ισχυρές πολιτικές για τις πόλεις. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το συμμερίζονται ε, πολλές χώρες μέλη. Υπάρχουν τα θέματα της επικουρικότητας εδώ και θα πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί τους. Αν δείτε πώς οι δήμαρχοι βλέπουν το θέμα, πιστεύουν οι δήμαρχοι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων για να μπορέσουμε να ε, μοιραστούμε τις γνώσεις μας, τις βέλτιστες πρακτικές προς το καλό των πολιτών και το καλό του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ζήλε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας κύριε Σεύκοβιτς. Από πλευράς της πολιτικής μας ομάδας θα θέλαμε να έχουμε μια σωστή συνεργασία μαζί σας. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε ε, ανησυχίες για τους λεγόμενους διαδρόμους του Connecting Europe. Ε, ε επίσης η συμμετοχή κοινοτική σε τέτοια προγράμματα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ε, οι κανόνες λένε ότι μέχρι το τέλος του 2016, εφόσον δεν συνεχιστούν ορισμένα προγράμματα, θα πρέπει να εφαρμόσει την αρχή του ε, χρησιμοποίησε τις πιστώσεις ή χάσε τις πιστώσεις. Οπότε τι θα κάνετε. Πολλές αποφάσεις μερικές φορές ε, εφαρμόζονται μόνο σε μία χώρα μέλος ε, κάτι το οποίο φυσικά δεν ε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το Connecting Europe λοιπόν θα πρέπει να αφορά πολλές χώρες κάθε φορά. Τώρα, οι υπερτήσεις στην πολιτική αεροπορία. Στα πλαίσια της κρίσης με την ε, Ρωσία κάποιες, ε, κάποιοι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την, ε, τον, σι, τον σιβηρικό εναέριο χώρο, λέει ο ομιλητής. Λοιπόν, η Ρωσία εδώ θα πρέπει ε, να σταματήσει ίσως να εισπράττει χρήματα από τους Ευρωπαίους αερομεταφορείς σε αυτή την περίπτωση. τι μέτρα, τι αντίμετρα θα έλεγα καλύτερα ε, σκοπεύετε να λάβετε εις βάρος της Ρωσίας γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Ζήλε για τις δύο ερωτήσεις σας. Ξεκινώντας με τους διαδρόμους του Connecting Europe. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη σχετικά με την δυνατότητα απορρόφησης των πιστώσεων. Είναι αλήθεια ότι το 2016 θα είναι μια κρίσιμη χρονικά στιγμή και θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και να δείξουμε ότι ε, ε, το εννοούμε αυτό το οποίο λέμε. Εάν φανεί ότι ε, δεν έχουν σεβαστεί κάποιοι εμπλεκόμενοι ε, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, τότε το θέμα της χρηματοδότησης με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τεθεί. Ήδη έχουμε περάσει ε, σε διαφορετικό πλέον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα έπρεπε να έχουν γίνει εν τω μεταξύ όλες οι αλλαγές που θα διασφαλίσουν την αύξηση της απορροφητικότητας από τα κράτη-μέλη και ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή use it or lose it. Ε, βέβαια πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα κρατημέλη γιατί μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να ε, εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θα τα εξετάσουμε αυτά προσεκτικά και θα τους δώσουμε με δίκαιο τρόπο μια προειδοποίηση. Κοιτάξτε, αν δεν τα χρησιμοποιήσετε τώρα κινδυνεύετε να τα χάσετε. Όλοι ελέγχουν εδώ και οι ελεγχόμενοι είναι αυτοί και ελέγχοντες είμαστε εμείς αλλά και εσείς σαν κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί λοιπόν σε σχέση με όλα αυτά και νομίζω ότι με την στήριξή σας θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα για την υπέρπτυση στη Σιβηρία. Ξέρετε ότι οι σχέσεις μας με την Ρωσία είναι ιδιαίτερω περίπλοκες, όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά και στον τομέα των οικονομικών και τις μεταφορές. Θα σταθώ στο θέμα των υπερπτήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε για πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις. Η τελευταία υπόσχεση των Ρώσων είναι ότι εφόσον μπούμε στον ΠΟΕ θα καταργήσουμε τα τέλη αυτά, τη τέλη υπέρπτυσης και δεν θα τα χρεώνουμε πλέον. Ε, μέχρι τώρα όμως οι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς πληρώνουν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά σαν επιδότηση ε, των ρωσικών αερογραμμών οι οποίες εταιρείε οι ρωσικές κάνουν τα ίδια δρομολόγια με τις δικές μας. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Κανονικά θα έπρεπε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Αυτό ελπίζω και θα εργαστώ γι' αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει ε, καλό να είναι οι Ευρωπαίοι να έχουν μία φωνή απέναντι στη ρωσική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει να υπάρξει μια συμφωνία για την υπέρκτηση της Σιβηρίας γιατί τα τέλη τα οποία εισπράττουν είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με τους διεθνείς κανόνες. Η κυρία από την ομάδα των φιλελευθέρων καλώ ήρθατε κύριε υποψήφια. Περιμένω τις απαντήσεις σας για τις ερωτήσεις που θα σας διατυπώσω. Θα ήθελα να επικεντρωθώ όπως και εσείς στο μεγαλύτερο μέρος στην αρχή της εκθέσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο των μεταφορών που βεβαίω και όλοι επιθυμούμε και ιδιαίτερα θα ήθελα να βάλω έμφαση στο χώρο των θαλασσίων μεταφορών αναφερθήκατε στη σημασία των λιμένων και ιδιαίτερα αυτό που με ικανοποίησε ήταν αυτό το οποίο ε, αναφέρατε για τις εσωτερικές πρώτες οδούς και τη σημασία τους που μπορούν να σημάνουν και αποσυμφόρηση των οδικών μεταφορών και την ενίσχυση βέβαια των θαλασσιών μεταφορών. Αυτό πρέπει να μπει μέσα στι θαλασσιέ μεταφορέ, γιατί έχουμε συζητήσει για ένα ε, δίκτυο των σιδηροδρόμων. Πρέπει να κοιτάξουμε και τι θαλάσσιε μεταφορέ, κυρίω τι εσωτερικέ πλωτέ οδού, όπου μα είπατε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό ακόμα που δεν έχει αξιοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξή θα πρέπει να αναπτυχθούν, δηλαδή να, βάλουμε πιο, να χτίσουμε πιο ψηλές γέφυρες, να σκάψουμε, να ανοίξουμε όχθες ε, σε ορισμένες περιοχές όπως και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Αυτό πώς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση, επί παραδείγματι... Το ζήτημα της ε, αντιδράσεως πολιτών ως προς την ε, διάνοιξη ε, πλωτών οδών στον Δούναβη ή στον Έλβα ακόμα έχουμε ε, δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας. Πώς μπορείτε λοιπόν να ε, οθήσετε τα κράτη-μέλη σε μια πιο καλή συνεργασία στον τομέα αυτών. Παρακαλώ, απάντηση. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για την ερώτησή σας. Έχετε πολύ το δίκαιο ότι δυστυχώς οι εσωτερικές πλωτές οδοί και οι μεταφορές αυτές έχουν παραμεληθεί κάπως. Και λόγος ήταν ότι ο στόλος ήταν παλαιωμένος, επαρχαιωμένος, δεν είχαν σωστή συντήρηση, εσωτερικές πλωτές οδοί και ότι ήταν πολύ κατακαιρματισμένος ο κλάδος, κυρίως με πολύ μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακές ακόμη μικροεπιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, δυνατούν να κάνουν πραγματικά μεγάλες επενδύσεις και να βοηθήσουν έτσι στην ε, μεγέθυνση του κλάδου πέρα από αυτή την πολύ περιορισμένη κλίμακα. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά βλέπω το, τα όσα έχουν γίνει και πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν πολλά στην τόσο υποσχόμενη αυτή ε, βιομηχανία στον κλάδο αυτόν τον τόσο υποσχόμενο και οικολογικά. Αν δει κανεί δηλαδή πόσα μεταφορά μπορούμε να φορτώσουμε πάνω σε μια μαούνα ή τι είδου εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να έχει σε σχέση με άλλων τύπων μεταφορέ, αλλά και τι είδου δυνατότητε προσφορά ε, διασυνδέσεων μεταξύ λιμένων μπορεί να σημάνουν αυτέ οι εσωτερικέ πλωτέ οδοί. Βλέπουμε ότι έχει τεράστιο δυναμικό αυτό ο κλάδο. Εάν λοιπόν με στηρίξετε και με βοηθήσετε στην υπόθεση αυτή, εγώ θα ήθελα να αξιοποιήσω το πρόγραμμα Ναϊάδες ώστε να βοηθήσω στην ανοικοδόμηση του κλάδου των εσωτερικών πλωτών οδών, ε, να βοηθήσω στην ανακαίνιση του κλάδου των πλοίων, στον ανασχεδιασμό κατά τρόπο οικολογικό και σύγχρονο των πλωτών οδών, κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης μορφής εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Και βεβαίως θα χρειαστεί και η στήριξη και η εντατική συνεργασία των κρατών μελών για την διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου πλοηγημότητας ε, στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ξέρετε ότι η πατρίδα μου, ιδιαίτερη η Μπρατισλάβα, πάνω στο Δούναβι, μου επιτρέπει να γνωρίζω πολύ καλά τι είδους προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και σε σχέση με τα γειτονικά κράτη. Ε, χρειάζεται λοιπόν πρόοδος οπωσδήποτε στο τομέα αυτόν. Με ενθαρρύνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πλοηγιμότητα του ε, Δούναβι έλαβε ιδιαίτερη σημασία στην ε, τοποθέτηση των κρατών της στρατηγικής για το Δούναβη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, είπαν ότι υπάρχει δυναμικό, θέλουν να δώσουν νέες δυνατότητες και στην περιφέρεια και στις σταστικά κέντρα και τις μικρότερες πόλεις που βρίσκονται πάνω στον Δούναβη και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε έτσι να καθησυχάσουμε και τους πολίτες ως προς τα προβλήματα που τους απασχολούν, δίνοντάς τους ότι υπάρχει δυναμικό, ένα δυναμικό το οποίο μπορούμε αναζωογονώντας αυτές τις οδούς και αυτόν τον τρόπο μεταφοράς να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα και τις περιφέρειες και τις πόλεις. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε και πρέπει να πράξουμε. Ευχαριστώ. Μαρία Κίλαρ. Κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε. Κύριε Σεύκοβιτς. θα έχω να σας θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτον για τις συνθήκες εργασίας. Όταν έχουμε όλο και μεγαλύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση στις αγορές μεταφορών και φαίνεται ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών κινδυνεύουν να μειωθούν κάτι το οποίο θα θίξει την βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιταχύνει την υποβάθμιση της ευρωπαϊκής πείρας, γνώσης και πείρας και την ύπαρξη <clears throat> εργαζόμενων στον τομέα μεταφορών που έχουν αφοσίωση στον τομέα αυτό. Ιδίως στην ε, αεροπορία οι λεγόμενες εταιρείε χαμηλού κόστους παίζουν κορώνα γράμματα την ασφάλεια και εφαρμόζουν συνθήκε εργασία όλο και χειρότερε. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τι ασφαλεί συνθήκε εργασία και ένα τρόπο εργασίας που αποτρέπει το κοινωνικό dumping. Ποια είναι τα σχέδιά σας επίσης για τους στόχους εκπομπών και ε, ψηφιακή ατζέντα. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ε, οικονομική ανάκαμψη στον τομέα των μεταφορών και, θα και πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ευμάρεια των πολιτών της. Η ψηφιοποίηση, η ψηφιακή ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και βοηθάει και σε θέματα και σε λύσεις προβλημάτων επιμελητίας. Είναι όμως ακόμα στα γενοφάσια της αυτή η διαδικασία στον τομέα μεταφορών, αλλά πιστεύουμε ότι χάρη στην ε, χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα ανοίξουν πολλές δυνατότητες. Φαίνεται όμως ότι οι ανταγωνιστές μας, οι ΗΠΑ, η Κίνα και άλλες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο τις ψηφιακές δυνατότητες από εμά. Ελπίζω θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και εμείς στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρόμους χωρίς κοινωνικό ντάμπινγκ. Πώς θα προωθήσετε λοιπόν τον τομέα μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρησιμοποιήσει περισσότερο τις ψηφιακές τεχνολογίες για να γίνει και πρώτοπόρο ο τομέας αυτός σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός διαλειτουργικού και βιώσιμου χώρου μεταφορών. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, έχετε το λόγο, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη και το χρόνο, γιατί το ερώτημα ήταν πράγματι μακροσκελές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, <clears throat> συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε η αξιότιμη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δείτε τους ε, οδηγούς θα χρειαστούμε χιλιάδες οδηγούς επιπλέον στην Γερμανία και στην Ολλανδία. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί από τους ε, μηχανοδηγούς των τρένων θα αποσυρθούν, θα πάρουν σύνταξη και θα χάσουμε την μεγάλη τους γνώση. Έχουμε χιλιάδες ναύτες από τις Φιλιππίνες στην ναυτιλία μας γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε κίντρα στην ε, νέα γενιά που είναι η πιο άνεργη νέα γενιά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να πάρει αυτές τις θέσεις εργασίας και να εργαστεί στον ε, ναυτιλιακό τομέα, στις μεταφορές. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να αλλάξουμε την αντίληψη που έχουμε για τις μεταφορές. Θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα και να παρουσιάσουμε το τομέα αυτό σαν ένα εργαλείο εξυγχρονισμού, σαν ένα οικονομικό κλάδος όπου μπορεί πράγματι κανείς να χρησιμοποιήσει υψηλές τεχνολογίες. Ένα τομέα όπου υπάρχει μια βιομηχανία που προετοιμάζει το μέλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό και στα σχολεία. Θα πρέπει να εργαστούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα για να βελτιώσουμε τις συνδίκες εργασίας. Γιατί πολλές φορές αυτό είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τι είδους ε, κοινωνικές συνθήκες εργασίας, τι είδους ε, αποδοχές θα έχει κάποιος ο οποίος θέλει να εργαστεί στον τομέα μεταφορών. Εάν θέλουμε να είναι ελκυστικό ο τομέα για να αντικαταστήσει αυτούς οι οποίοι θα ε, συνταξιοδοτηθούν μέσα στα 10-15 χρόνια, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Για τις ψηφιακές τεχνολογίες, εδώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ γρήγορη η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και κυρίως πιστεύω θα υπάρξει και μεγαλύτερη σύνδεση με τις τεχνολογίες του διαστήματος σχετικά. Η Κάρη Μαντέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν θέσω την ερώτησή μου θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εννέα μόνο γυναίκες εμείς ε, είχαμε κάνει τεράστιους αγώνες, αλλά εσείς ε, δεν φταίτε κύριε Σεύκοβιτς, οπότε εξ ονόματος των Πρασίνων σας, ε, σας καλωσορίζω. Και συνεχίζω στα γαλλικά, μιας και μιλάτε πολύ καλά. Η συμφωνία θα πρέπει να κλείσει, η συμφωνία 21, δηλαδή πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε και τη συνάντηση κορυφής για το κλίμα ε, παρόλα αυτά το θέμα των μεταφορών δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής για το κλίμα, ενώ είναι κατεπίγοντα τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά. Ε, έχετε ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τη συνάντηση αυτή κορυφής για το κλίμα. Η Επιτροπή είπε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία εμείς θεωρούμε άχρηστα όπως η συνδεση το Λιόν-Τωρίνο ε, είναι κάτι το οποίο έχει, θα αυξήσει το κόστος ε, άλλωστε και για τις μεταφορές πάρα πολύ ε, υψηλά. Έτσι κι αλλιώς έχουν υποεκτιμηθεί οι δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά 30% τουλάχιστον, ενώ υπάρχουν πολλά να γίνουν για την βελτίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές. Στη Γαλλία 8 εκατομμύρια Γάλλοι σαν παράδειγμα δεν έχουν πρόσβαση στις μεταφορές. Ε, ε, βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς χαρακτηρίζει και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Και γιατί το Συμβούλιο και η Επιτροπή αυτά τα λίγα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσουν για άχρηστους λόγους. Πώς μπορεί λοιπόν να χρηματοδοτεί αυτά τα άχρηστα προγράμματα όπως το Λιόν ρίνο, ενώ θα μπορούσε και στα πλαίσια του RTE να δαπανίσει καλύτερα τα χρήματα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην παρούσα φάση την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος αυτού, όπως επίσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πώς μπορεί λοιπόν από τη μία να σεβαστεί αυτό το 3% του ΑΕΠ που προβλέπεται από τις συνθήκες και από την άλλη ε, ε, τα προβλήματα, τα δημοσιονομικά που δημιουργούν τα σχέδια αυτά σε πολλές χώρες. Σας ευχαριστώ κυρία Ντέλη και για τα καλά σας λόγια στην αρχή της παρουσίασής σας. Αν μου επιτρέψετε τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί η ορολογία μου ε, σε σχέση με αυτούς τους νέους τομείς ε, είναι περιορισμένοι, αλλά συνεργαζόμενοι θα βελτιωθούν και οι γλωσσικές μου γνώσεις για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συνάντηση κορυφή στο Παρίσι για το κλίμα θα είναι ε, κρίσιμη. Ε, νομίζω ότι ακόμα και αν η Ευρώπη μπορεί πράγματι να κάνει περισσότερα από ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, ε, πάντα κάνουμε περισσότερα από τους άλλους ε, παγκόσμιους εταίρους μας, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλέον επιχειρήματα για να τους πείσουμε να πάρουν μέρος σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για να φροντίσουμε το κλίμα στον πλανήτη. Ο συνάδελφος Πότοτσεκ λέει ότι ο πλανήτης θα επιβιώσει των ανθρώπινων ενεργειών. Εμείς όμως θα επιβιώσουμε πάνω στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι απαιτείται να δείξουμε ότι είμαστε φιλόδοξοι και να πρέπει να έχουμε μια σφαιρική θα έλεγα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενθαρρύνθηκα όταν είδα πάρα πολλές προσωπικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες μέρες να δηλώνουν την αφοσίωσή τους προς τους στόχους αυτούς και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη συμμετοχή μας θετικά στο Παρίσι. Τώρα σχετικά με τα θέματα τα περιβαλλοντικά γενικότερα. Βλέπετε εδώ όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε για το περιβάλλον. Ε, ε, στρατηγική 2020, στόχοι 2020, στόχοι 2030. Ξέρω ότι θα είμαστε επιτυχείς σε πολλούς τομείς, ε, λιγότερο ή περισσότερο. Νομίζω ότι και στις μεταφορές μέσω κάποιων κανονισμών, μέσω της πίεσης της βιομηχανίας να είναι πιο αποδοτική ενεργειακά, να χρησιμοποιήσει νέους τύπους ε, κινητήρες, Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν βελτιώσει κάπως την κατάσταση. Οι στόχοι λοιπόν που έχουμε εδώ είναι δεσμευτικοί στόχοι όπως είπαμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε τις πιέσεις έτσι ώστε να μειωθεί η μόλυνση. Δεν έχω χρόνο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, λυπάμαι. Λούγκρεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Σεφκοβίτς που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω κάποιες ε, ε, σκέψεις, να εκφράσω κάποιες σκέψεις για το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, εν πολλής Αλλά από την άλλη με τρομάζει κιόλα. Από τότε που ήσασταν 18 δεν βλέπω να κάνατε ούτε μια μέρα χειρονακτική δουλειά. Τώρα έρχεται να, κάνετε, να αναλάβετε καθήκοντα σε μια πολύ ψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αποφάσει θα επηρεάζουν την ε, ζωή και τη δουλειά εκατομμυρίων πολιτών, που εργάζονται στις μεταφορές, χωρίς να έχετε την παραμικρή εμπειρία από το χώρο αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι εγώ ο Σουηδός δεν θα μπορέσω να, σου, να εξηγήσω στους, ε, στο εκλογικό σώμα, κυρίως όσους ψηφοφόρους προέρχονται από τις μεταφορές, ότι ήσασταν ο καλύτερος ψήφισε τον τομέα αυτόν, γιατί δεν έχετε την παραμικρή εμπειρία. Και δεν γνωρίζετε τα σοβαρά προβλήματα του τομέα μεγαλώσατε και ανδρωθήκατε μέσα σε ένα χώρο με υψηλές σπουδέ, με πολιτική δραστηριότητα, με απίστευτους μισθού, μισθούς σε σχέση με αυτούς που υποτίθεται ότι θα εκπροσωπήσετε. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα ε, δεν καταλαβαίνω πώς θα τους εκπροσωπήσετε λοιπόν. Και κύριε Σεύκοβιτς, το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι τεράστιο στον τομέα των μεταφορών. Ένα πρόβλημα το οποίο απορριθμίζει και αποδιαρθρώνει κάθε είδους ε, εταιρεία. Εμείς στην πατρίδα μου έχουμε για τις οδικές μεταφορές το πρόβλημα αλλοδαπών οδηγών φορτηγών, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν τις μεταφορές με τίμημα ε, τίμημα με το 1 τρίτο των δικών μας οδηγών. Κατοντάδες επιχειρήσεις μεταφορών έκλεισαν πέρυσι λόγω ακριβώς της απουσίας προστασίας εναντί αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού στη Σουηδία. Οι επιχειρήσει μα δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται σε όρου ισοδύναμου. Πώ μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε τέτοιου είδου ισότιμου όρου όταν το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι ένας, ένα, ένα είδο πλεονεκτήματο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για τα ευγενή σας λόγια για το βιογραφικό μου σημείωμα. Σας βεβαιώνω όμως ότι γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει χειρονακτική εργασία γιατί όταν ε, μεγάλωνα ε, ως νέος είχα όπως κάθε νέος ε, την ευκαιρία να εργάζομαι υποχρεωτικά τα καλά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάθε φοιτητή ήταν υποχρεωτικό να δουλεύει στα εργοστάσια. Το ίδιο συνέβη και όταν ήμουν μετά στη Ρωσία ως φοιτητή. Αυτή είναι μια εμπειρία που πολύ ευχαρίστω να μοιραστώ μαζί σας. Γνωρίζω λοιπόν πόσο σκληρή είναι αυτή η δουλειά και γνωρίζω με τι είδους στρες και άγχος δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερα δε στις οδικές μεταφορές το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι ασφαλώς ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ήθελα λοιπόν ε, να σημειώσω, όπως είπα και στις αρχικές μου παρεμβάσεις, αλλά με χαρά θα το τονίσω και πάλι, είναι ότι θέλω μαζί με σας να κοιτάξουμε εις βάθος και συνολικά το τι μπορεί να απλουστευθεί, το τι μπορεί να διευκρινιστεί ως προς τους κανόνες που εφαρμόζονται στις μεταφορές. Γιατί όσο πιο απλοί είναι οι κανόνες, όσο πιο ξεκάθαροι, τόσο πιο ευχερής και η ε, ε, επιβολή τους και φαντάζομαι ότι θα μας στηρίξουν και οι κυβερνήσεις και οι αρχές που καλούνται να τηρήσουν και να εφαρμόσουν κανόνες αυτούς, έτσι ώστε να έχουμε απλούς κανόνες, σαφείς κανόνες, δίκαιους, ισοδίκαιους κανόνες και βέβαια από εκεί και πέρα θα πρέπει οι εθνικές αρχές να μεριμνήσουν για την επιβολή τους. Τώρα για το πρόβλημα συγκεκριμένα των οδικών μεταφορών που αναφέρατε, εγώ πάλι μαζί με εσά. Θα είμαι διατεθειμένο να προτείνω στου κοινωνικού εταίρου την βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου και την αναζήτηση μια λύση, η οποία παραδείγματι θα σήμαινε ε, το να μην χρειάζεται πάντοτε η παρέμβαση ε, στα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στον χώρο των οδικών μεταφορών. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ απλό αυτό ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ε, εφόσον βέβαια οι κανόνες είναι σαφείς και ευχερείς στην εφαρμογή τους για να έχουμε ένα σαφή και ε, σταθερό χώρο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο. Τρία λεπτά ερώτηση και απάντηση πάντα και οι γραμμές είναι μία, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Παρακαλώ τηρήστε τον καρόνα αυτόν. Όσο πιο σαφείς είστε και σύντομοι τόσο πιο διεξοδικά μπορεί να απαντήσει ο υποψήφιος επίτροπος. Ο κύριος Κόχ είναι τώρα επόμενος. Είναι πίσω σας κύριε Σέρκοβιτς, μην ψάχνετε στην αίθουσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεύκοβιτ, κάθομαι πίσω σα και ελπίζω μετά την ακρόαση να μπορώ να σταθώ στο πλευρό σα και να σα στηρίξω κι εγώ με την, με ψήφο μου. Έχουμε λοιπόν ε, να μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και με πάρα πολλά προβλήματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει τη Λευκή Βίβλο με προγράμματα για τις μεταφορές, τις οδικές μεταφορές ε, και εδώ το θέμα μας είναι η ασφάλεια βέβαια και χιλιάδες νεκρών στους δρόμους ε, της Ευρώπης. Ε, ο στόχος λοιπόν της Λευκής Βίβλου ήταν να περιοριστούν ε, οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα. Εγώ ήμουν εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ήρθε το θέμα στην έκθεση και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είδους συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε εφόσον επιβεβαιωθείτε στη θέση του Επιτρόπου προκειμένου να εκμηδενίσετε τον κίνδυνο των τροχαίων δυστυχημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόχ για την ερώτησή σας. Έχει τεράστια σημασία πιστεύω για εκατοντάδες χιλιάδων Ευρωπαίους όχι μόνο 26.000 νεκροί πέρσι, 250.000 σοβαρά τραυματίες επίσης καταγράφηκαν σε ε, τροχέα το 2013 και μπορεί να λέμε ότι είναι η πιο ασφαλής, ο πιο ασφαλής χώρος των μεταφορών η Ευρώπη, αλλά σε απόλυτους όρους τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτα υψηλά. Αλλά να δούμε λίγο τα στοιχεία. Το 2014 παρότι είχαμε πολύ σταθερή μειωτική τάση, ως προς τον αριθμό των θυμάτων των τροχαίων τα τελευταία χρόνια με μείωση κατά 18% βλέπουμε ότι το 2014 μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφρά αύξηση των στατιστικών στοιχείων. Θα πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Υπάρχουν λόγοι όπως η παραδείγματι πολύ ε, μακρύς ή άλλοι παράγοντες. Ε, πάντως είναι ανησυχητικά τα στοιχεία. Και ήδη αυτό που ε, έχει φέρει καρπούς είναι η αναζήτηση των λόγων και βέβαια πρέπει από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αφενός μεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία ε, η σχετική με την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, ε, επί παραδείγματι οδηγοί οι οποίοι μέχρι τώρα οδηγούσαν ε, κατά τρόπο επικίνδυνο επειδή βρίσκονταν έξω από τα σύνορα τα οδικά της χώρας τους, τώρα θα κινδυνεύουν με πρόστιμο και εφόσον έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ξένες χώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Μπορούμε επίσης να δούμε άλλους τρόπους να μειώσουμε τα σοβαρά, τους σοβαρούς τραυματισμούς που προκύπτουν από τα τροχέα ε, και πολλά άλλα θετικά μέτρα που μπορούμε να αναλάβουμε στα αστικά κέντρα με νέες ε, προσεγγίσεις και λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν ε, ακόμη και αυτόν που έχει εμπλεκεί, αυτόν έχει εμπλεκεί κάποιο ένα ατύχημα, να βοηθήσουν στην ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο κύριος Σασόλη έχει το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον υποψήφιο επίτροπο να του θυμίσω μάλλον ότι στην τελευταία συνάντηση που πήραν μέρος οι συντονιστές της Επιτροπής Μεταφορών και οι εισηγητές για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο ε, συζητήθηκε να δοθεί στο Κοινοβούλιο ε, η εντολή διαπραγμάτευσης ε, και του τεχνικού πυλώνα αλλά και του πολιτικού πυλώνα. Πιστεύετε κύριε Επίτροπε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πιστεύετε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον προηγούμενο Φεβρουάριο μπορεί να αντιπροσωπεύσει την σωστή διαπραγματευτική βάση για τους επερχόμενους τριμερείς διαλόγους. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να υιοθετήσει το 15 την αλλαγή του κανονισμού ΕΑΣΑ, εάν σε αυτή την περίπτωση είναι καταφατική η, απόφαση, η απάντησή σας, Πώς θα ξεκινήσετε ε, τις διαπραγματεύσεις αυτές για το ΣΥΝ 2. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ κύριε σας όλοι για τις ερωτήσεις σας. Είναι θέματα τα οποία πράγματι βρίσκονται στο τραπέζι το νομοθετικό στην παρούσα φάση και είναι ένα θέμα στο οποίο καλούμε εφόσον πρόταθω να ασχοληθώ γρήγορα. Η Ιταλική Προεδρία υποστηρίζει ιδιαίτερα το πακέτο το σιροδρομικό. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην διαπραγμάτευση. Έχουν υπάρξει, ε, προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση των αρμόδιων Υπουργών Μεταφορών για το θέμα αυτό και οι Υπουργοί θα πρέπει ε, να στηρίξουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την σοφή κατεμέ, τη συνοχή αυτών των προτάσεων σε ένα πακέτο. Έχουν υπάρξει βήματα προόδου σε επίπεδο τεχνικό. Βέβαια υπάρχουν τεχνικά προβλήματα τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδι για την σιδηροδρομική βιομηχανία. Αλλά θα πρέπει και στο πολιτικό κομμάτι να κάνουμε βήματα προόδου η ανάπτυξη μέσων εμπιστοσύνης, δημιουργίας εμπιστοσύνης, κλίματος εμπιστοσύνης νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε σωστές λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία της Επιτροπής σας και του συνόλου της Ολομέλειάς σας. Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε και με την αναθεώρηση του ΕΑΣΑ ε, όχι ότι δεν κάνει πολύ καλή δουλειά η άσα. υπάρχουν εξαιρετικά άτομα εκεί που κρατούν την ασφάλεια στις πτήσεις στο ίδιο επίπεδο με τη ΣΥΠΑ. Θα θέλαμε όμως να, να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και η πρόοδος στο πακέτο ΣΥΝ2 θα δώσει δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, αναφερθήκατε ήδη στον, στους εθέρε εθέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά πρέπει και τα κράτη-μέλη να πιστούν να σταματήσουν την στεναρή αντίδραση που έχουν δείξει για να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα των ενιαίων εθέρων. Πρέπει για να γίνει αυτό πραγματικότητα να εφαρμοστεί το ΣΕΣΑΡ. Το ερώτημα είναι πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και του σχεδίου ΣΕΣΑΡ και πάλι είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον εναέριο έλεγχο πάνω από την Ευρώπη. Ένα ακόμα <clears throat> ερώτημα για το πρόγραμμα Έγνος καλύπτει το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου ως διαστημικό πρόγραμμα. Τότε θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τις ε, διαδικασίες προσγείωσης στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πότε νομίζετε ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα έγνωση από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και επίσης για, το, για τις κοινωνικές συνθήκες τι άποψη έχετε για τα πρόστιμα που χρειάστηκε να πληρώσουν οι οδηγοί φορτηγών που έχουν ξεπεράσει το χρόνο που περνάνε μάλλον το χρόνο ανάπαυσή του στι καμπίνε των φορτηγών, παραδείγματο χάρη αυτό στη Γαλλία. Και αν θέλετε, μπορώ να, να σα πω πώ ήταν τα πράγματα και στη δική μου χώρα πριν πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαϊνέσκου. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό γιατί είσαστε πραγματικά εμπειρογνώμων, υπήρξατε υπουργό μεταφορών και είστε και μηχανολόγος. Το πρώτο ερώτημά μου, η ερώτημά σας, συγγνώμη. Δεν μπορώ να μην πω ότι νιώθω μεγάλη ματέωση για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος για τα λεγόμενα block εθέρων. Είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε ένα σύστημα που θα μοιάζει με το σύστημα των ΗΠΑ που είναι ενίος ο ενάριο χώρος. Ελπίζω όμως ότι αυτά τα εννέα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου θα μπορέσουν να γίνουν, νόμιζω θα γίνουν πραγματικότητα, αλλά ούτε και αυτό έχει καταστεί δυνατό. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για μένα για αυτό το γεγονός. Αν θέλουμε να χάνουμε 5 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επειδή δεν θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα, είναι πραγματικά απώλεια χρημάτων. Το ΣΕΖΑ θα μπορούσε να βοηθήσει γιατί και εξάλλου έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους ανταγωνιστές μας. Ξέρουμε ότι κάποιες ασιατικές χώρες έχουν ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το σχέδιο Σέζαν. Είναι πιο <clears throat> αποτελεσματικό, επιτρέπει τα αεροπλάνα να πετούν πιο κοντά το ένα το άλλο, να υπάρχει καλύτερη χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου και εξασφαλίζει και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αεροδρόμια. Για να κλείσω λοιπόν αυτό το σημείο, θα προχωρήσω στο διορισμό ενός μάνατζερ ανάπτυξης για το ΣΕΣΑΡ που ελπίζω ότι θα προωθήσει σε πραγματική εφαρμογή αυτό το σχέδιο στην Ευρώπη και συγγνώμη τελείωσε ο χρόνος μου. Ναι, φταίει η ερώτηση που ήταν πάρα πολύ μακροσκελής. Κύριε Ταπαρντέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το δικό μου ερώτημα είναι πιο άμεσο και πιο συγκεκριμένο. Αφορά το τέταρτο σιδηροδρομικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τον πολιτικό πυλόν αυτού του πακέτου. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με την πρόθεση του τομέα αυτού. <clears throat> Υποστηρίζετε την αρχή του, του ανταγωνισμού και για τον τουρισμό. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό το τμήμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ μεταφορών και τουρισμού. Υπάρχουν πολλές ελκυστικές περιοχές για τον τουρισμό στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη προσβασιμότητα όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί, Γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Τι στρατηγική θεωρείτε ότι, να, ότι πρέπει να εφαρμοστεί για να υπάρξει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στις περιοχές αυτές που έχουν μεγάλο δυναμικό για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε ότι ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ΑΕΤ της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και είναι απαραίτητε μεταφορέ για τον τουρισμό. Τρίτο ερώτημα. Τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τη Ρουμανία, τη χώρα από την οποία προέρχομαι εγώ. Οι χώρε αυτέ είναι συνδεδεμένες με χώρες έξω από την Ευρώπη, με την Κίνα, τη Ρωσία, την Αποανατολή, τι στρατηγικέ θα πρέπει να εφαρμοστεί στι χώρε αυτέ για να αναπτύξουν περαιτέρω στα σύνορά του τι υποδομέ του μεταφορών. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση με του ανατολικού μα ε, γείτονε, όχι μόνο σε επίπεδο μεταφορών, αλλά σε και επίπεδο οικονομικών σχέσεων. Οι μεταφορέ λοιπόν με τι υποδομέ και την ε, λειτουργία τη είναι ένα από του πυλώνε Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνοντα. Πρέπει να πω ότι είναι λίγες οι γυναίκες που είναι ε, <clears throat> επίτροποι, αλλά έχουμε πολλές γυναίκες στην Επιτροπή Μεταφορών και αυτό είναι θετικό. Μένει ένα λεπτό μονάχα για τον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εάν δεν λάβετε όλες τις απαντήσεις που περιμένετε θα είναι δική σας ευθύνη διότι δεν ε, αφήσατε αρκετό χρόνο, μιλήσατε πάρα πολύ ωραία. Όπως είχα πει, ούκεν το πολλό το F και ως εκ τούτου θα δώσω στον ε, Επίτροπο το λόγο για όσο χρόνο περισσεύει τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη διμερή συνάντηση για όλες αυτές τις ερωτήσεις από ό,τι διαπιστώνω. Πάντως θα ήθελα να πω ότι για το πακέτο για τους σιδηροδρόμους θα πρέπει να βρούμε μια λύση αποδεκτή για την πλειονότητα των ε, κρατών μελών και βέβαια την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με λύσεις ε, διαφορετικές και ποικίλε τις οποίες είμαι τεθειμένος να εξετάσω στο σύνολό τους, αλλά πάνω απ' όλα έχει σημασία να εξασφαλιστεί πρόοδος. Θα πρέπει επίση να αναπτύξουμε τι δυνατότητε που μα δίνουν τα ερθωτικά ταμεία και εδώ έχουν ευθύνη τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε πόσο ποιοτικέ ε, υποδομέ μεταφορών μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζει κανεί ότι θα ταξιδέψει κάπου με τρόπο ασφαλή και ευχερή και μπορούμε χάρη στα ερωτικά ταμεία να προωθήσουμε και τα τουριστικά αξιοθέατα στις ε, χώρες μας. Αυτό θα είναι πολύ σοβαρή επένδυση για το μέλλον, ο Πρόεδρος. Τέρμα, θα πρέπει δυστυχώς για να είμαι δίκαιος προς όλους να σας διακόψω. Δεν είναι δική σας ευθύνη βέβαια. Α, ο κύριος Κλούν έχει το λόγο. Κυρία Κλούν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα ίσως να βοηθήσω με τις ερωτήσεις της συνάδελφο για να πάρουμε τις απαντήσεις. Ε, θα θέλαμε σε σχέση με τις απομονωμένες και τις πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές της ε, περιφέρειας ή το υπαίθρου της Ευρώπης να μιλήσουμε όταν υπάρχουν εκεί αεροδρόμια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν βέβαια και για την πρόσβαση σε τουριστικά αξιοθέματα κτλ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν στα περιφερειακά αεροδρόμια που κινδυνεύουν με κλείσιμο να διαφυλαχθούν. Οι κρατικές ενισχύσεις και οι σχετικοί κανόνες πρέπει να αξιολογηθούν βεβαίως, αλλά δεν θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα προβλήματα, όπως αναφέρω, των περιφερειακών, των απομονωμένων και των ισοτικών περιοχών της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι τοπικές περιφερειακές αεροπορικές συνδέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως και τα περιφερειακά αεροδρόμια αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ικανότητα, η χωρητικότητα των αεροδρομίων αυτών στην Ευρώπη και άμα δείτε και τη γειτονιά μας, βλέπετε ότι η γειτονιά μας προχωρά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν δείτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης που σύντομα θα μπορεί να υποδέχεται 140-150 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Μα βλέπετε τι γίνεται στο Ντουμπάι, όπου αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει στα 160 εκατομμύρια επιβάτες τον ε, χρόνο, ενώ στο Χήθρο έχουμε μονάχα 70 εκατομμύρια το maximum, <clears throat> βλέπετε ότι οι εξελίξεις στην ε, Μέση Ανατολή και στη γειτονιά μας είναι τόσο έντονες που θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αεροδρόμια μας και πώς αντιμετωπίζουμε τις αεναερίες μεταφορές ως σύνολο. Φυσικά είναι σημαντική η αύξηση της αποδοτικότητας στον αέρα και στα αεροδρόμια πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή λύση για να αναπτύξουμε το πακέτο για την χωρητικότητα των αεροδρομίων. Πιστεύουμε ότι αν, εφαρμόσουμε τις, αν εφαρμοστούν οι προτάσεις που έχουμε κάνει και ξέρω βέβαια και ποια είναι τα προβλήματα που εμπεριέχουν, μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα των αεροπολικών των αεροδρομίων στην Ευρώπη κατά 20 εκατομμύρια επιβάσεις το χρόνο χωρίς να προσθέσουμε ούτε ένα διάδρομο απογείωσης προσγείωσης. Πρέπει λοιπόν να εγκριθεί αυτό το πακέτο σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις, νομίζω ότι οι κατευθυντέριες γραμμές για τις επιδοτήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα είναι πολύ θετικές. Είναι καλό που ότι τις έχουμε. Γιατί ξέρω ότι αργότερα θα συζητήσετε και την κατάσταση των λιμένων και πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια τουλάχιστον έχουμε καλούς κανόνες για να αξιολογούμε τις κρατικές επιδοτήσεις και αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσω μαζί με την κυρία Βέσταγκερ, τη συνάδελφό μου που θα είναι αρμόδια για τις, ελπίζω για τα θέματα ανταγωνισμού και που θα καλύπτει και τις μεταφορές. Ο κύριος Πορέμπα έχει τώρα το λόγο, ο είναι και αυτός πίσω σας. Κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα δύο πράγματα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε. Σχετικά με το δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη. Καταρχάς, ο δικός άξον Βία Καρπάτια που ε, εκινεί στην Λιθουανία και περνά από την Σλοβακία, την Τσεχία και καταλήγει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν συμπεριλήφθη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αλλά υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία εδώ από τις περιφέρειες αυτές έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί και στα πλαίσια του Connecting Europe αν είναι δυνατόν. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Θα βοηθήσετε έτσι ώστε να δοθεί στο μέλλον μια επιτυχής κατάληξη σε αυτή την προσπάθεια γιατί αυτός ο οδικός άξον είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής. Τώρα, συνοπτικά οι σιδηρόδρομοι ε, τους οποίους ε, θα χαράξει η Ρωσική Ομοσπονδία μέσω Σλοβακίας και Αυστρίας. European funds. Thank you. Thank you very much, Mr. for... <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πορέμπα και για τις δύο ερωτήσεις σας. Σχετικά με την Βία Καρπάτια, είναι αλήθεια ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στα TENS αλλά έχει συμπεριληφθεί στο λεγόμενο συνολικό δίκτυο, ολοκληρωμένο καλύτερα δίκτυο το, και αυτό δείχνει την σημασία που έχει η ανάπτυξη των, των μεταφορών στην Ευρώπη σε αυτή την περιοχή ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε ε, και τα ταμεία συνοχής τα οποία έχουν στην δυνατότητά τους οι χώρες αυτές γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα κριτήριο που λέει ότι αν σε αυτό το συνολικό δίκτυο υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ε, ε, ευρύτερης ευρωπαϊκής σημασίας και διαμεθοριακά μεγάλης σημασίας. Νομίζω λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε στην Ανατολική Ευρώπη είναι η ποιότητα του προγράμματος ή η δυνατότητα απορρόφησης των πιστώσεων που είναι διαθέσιμα για τα διαφορετικά ταμεία στις χώρες αυτές και η ταχύτητα γενικά σχεδίασης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι αν δεν υπάρξει αυτή η προσπάθεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής. Μιλήσατε για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τομείς των μεταφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει σε αυτά και είχαμε και μια συμφωνία διακομματική γύρω από αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2012 και του 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών και αυτών με μειωμένη κινητικότητα που θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά σε σχέση και με ε, τα δρομολόγια και στις αερομεταφορές και θα πρέπει να μην υπάρχουν εξαιρέσεις από την ευθύνη των αερομεταφορέων στην περίπτωση καθυστερήσεων για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Σαν παράδειγμα θα το πω ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα στον τομέα των δικαιωμάτων αλλά δυστυχώς πολλά μένει να γίνουν και το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει επίσης και για τα νυχτερινά τρένα. Uh, τα δικαιώματα των επιβατών έχετε ε, πολύ σωστά που αναφέρεστε στον όρο «We've come a long way», διανύσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου Πράγματι έχετε πιέσει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών να είναι σε ε, εξέχουσα θέση. Το επόμενο βήμα τώρα. Το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πόσο τα δικαιώματα των ε, ε, επιβατών θα ενταχθούν στα πλαίσια των νέων διατροπικών μορφών μεταφορών. Αν αλλάζει κανείς σαν παράδειγμα μέσο από τρένο σε αεροπλάνο ή σε πλοίο κτλ. θα πρέπει να διατηρείται ο σεβασμός των δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο με απασχολεί ε, βλέπουμε ότι μόνο το 5% των επιβατών αυτή τη στιγμή έχουν αποζημιωθεί σαν παράδειγμα στην περίπτωση που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ένα σωστό μηχανισμό επιβολής και γιατί είναι περίπλοκοι οι κανόνες, αλλά και γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε το σεβασμό των κανόνων αυτών στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε τις παραβάσεις αυτές, τις καθυστερήσεις αυτές, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν πού πρέπει να προσφύγουν και να μην εξαρτώνται μόνο από την τοπική δικαιοσύνη για να αποζημιωθούν για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Για τους επιβάτες μειωμένης κινητικότητας, εδώ θα συνεργαστώ με την κυρία Τίσεν, ε, για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας που θα δίδει με το νόμο την εγγύηση ότι οι επιβάτες αυτοί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους ε, επιβάτες. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στις πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές ακόμα και αυτοί που έχουν προβλήματα όρασης μέσω των smartphones, των εφιών κινητών τηλεφώνων. κυρία Τσασκούν Μπιλμπάου Μπαραντίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς. Το τέταρτο συνδρομικό πακέτο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ευδοκίμησε το τρίτο το να υπάρχει μια νέα διακυβέρνηση στις μεταφορές που ξεπερνάει τα ιστορικά μονοπόλια και τις τα εθνικά στεγανά. Θέλετε να το κάνετε αυτό. Υπάρχει μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο για τις έξι εκθέσεις, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία. Θίγει τις εταιρείε που θέλουν ασφάλεια δικαίου και αυξάνει το κόστος της γραφειοκρατίας. Αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, ε, είσαστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην οδηγία στην εφαρμογή τη οδηγία για τη διαλειτουργικότητα χωρί πολιτική υποστήριξη. Θα κάνετε μελέτε για να δείτε ποιε είναι οι συνέπειε που θα προκύψουν από το τέταρτο πακέτο για τις επενδύσει και την απασχόληση. Τι θα γίνει αν δεν εγκριθεί για αυτά που ανέφερα και για την καινοτομία και την διαλειτουργικότητα στο σιδηροδρόμο. Και τέταρτον, πώ θα υποστηρίξετε το shift to rail, αυτό το κοινό εγχείρημα που είναι σημαντικό για του σιδηροδρόμου. Και τέλο, τι πιστεύετε για την διαχείριση, το, για την διάκριση μεταξύ διαχειριστών υποδομών και των αυτών που λειτουργούν τις ιδεοδομικές γραμμές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας, γιατί νομίζω ότι βρίσκονται στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων για το τέταρτο ιδεοδομικό πακέτο. Αν ήξερα όλες τις απαντήσεις για αυτά θα ήμασταν πολύ κοντά. Αλλά <clears throat> μπορώ να σας δώσω τη δική μου αίσθηση όπως βλέπω τώρα τα πράγματα. Η πρώτη προτεραιότητα για μένα είναι να διατηρηθεί ω σύνολο αυτό το πακέτο. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ καλά στα, έχουμε προχωρήσει καλά στα τεχνικά στοιχεία του πακέτου, αλλά θα ήταν κρίμα λόγω τη πρόοδου στο τεχνικό επίπεδο και των προβλημάτων που έχουμε στο πολιτικό επίπεδο, το επίπεδο διακυβέρνηση, να εγκαταλείψουμε αυτό το πακέτο. Για να είμαι ειλικρινή, δεν θέλω να έρθω να σα με ένα πέμπτο σιδηροδρομικό πακέτο. Θα είμαι πολύ ικανοποιημένο αν το τέταρτο πακέτο είναι το τελευταίο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν επιληθεί. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικά υποδείγματα. Έχουμε υποδείγματα που υπάρχει πλήρης ε, ε, διάκριση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών μεταφορών και του διαχειριστή των υποδομών, που έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο την απασχόληση στον ε, <clears throat> σιδηροδρομικό χώρο και, την, ε, και δυσκολίες για τις εταιρείες αυτές. Είμαι έτοιμος να ακούσω αυτές τις προτάσεις αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι η ισότητα ανταγωνισμού, η δημοσιονομική διαφάνεια και η κοινή κατανόηση ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος που θα εξασφαλίσει την ισότητα ανταγωνισμού για όλους τους συνδρομικούς φορείς και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βάλουμε σε νέες ράγες τον συνδρομικό τομέα στην Ευρώπη και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε και σε πέμπτο συνδεδομικό πακέτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφοι Επίτροπε. Ε, κανονικά θα πρέπει να μετατρέψουμε τις οικονομικές μεταφορές και να τις κάνουμε αποδοτικές ενεργειακά ε, και ε, εποφελείς για τις επιχειρήσεις και για τους επιβάτες δεν έχουν το ποσοστό στις μεταφορές συνολικά το οποίο τους αξίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια στη σωστή τους ανάπτυξη. Υπάρχει και αντίσταση από διάφορες χώρες που ε, εμένουν να κρατούν τις αρμοδιότητες τους γύρω από τη ρύθμιση των σιωδρομικών μεταφορών. Ε, με το άνοιγμα των εθνικών αγορών θα πρέπει να μην ε, παρεμποδίζουν ε, την είσοδο στην αγορά κάποιων εταιριών και δεν θα πρέπει να ενισχύουν τις παραδοσιακές ιοδρομικές εταιρείες που ελέγχουν και έχουν τα μονοπόλια. Και τι γίνεται με τις λεγόμενες ρήτρε αμοιβαιότητα στον τομέα των σιωδρομικών μεταφορών. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, είναι πεθεμητή. Νομίζω ότι ε, μου δίδεται τα επιχειρήματα για να προωθήσω και τα δύο τμήματα του πακέτου από κοινού. Δηλαδή απαιτείται πρόοδο στο τεχνικό κομμάτι, απαιτείται όμως και πρόοδος στον τομέα τον τεχνικό. Τα κράτη-μέλη και οι εταιρείες δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι δεν υπάρχει σωστός ανταγωνισμός και ότι υπάρχουν στρεβλώσεις εις βάρος τους σε κάποιες χώρες μπορεί να έχουν υπάρξει αναθέσεις ε, επιχειρηματικών σιωδρομικών δραστηριοτήτων χωρίς ε, δημόσιους διαγωνισμούς και διαδικασίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει και η απαιτούμενη διαφάνεια δημιουργείται η αίσθηση ότι τα χρήματα τα οποία δίδονται στις επιχειρήσεις τις ιοδρομικές για τη διαχείριση των υποδομών χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους θέσης. και χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για την εξαγορά επιχειρήσεων ανταγωνιστικών σε όμορες χώρες. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω της σωστής διαδικασίας διαφάνειας και ξεκάθαρων κανόνων. Έχω την ελπίδα ότι μετά από μια μεταβατική περίοδο η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερος μακρά θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι αν περάσουμε στην εφαρμογή των κανόνων γύρω από τις ρήτρες αμοιβαιότητας θα δημιουργήσουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί να ολοκληρώσουμε δηλαδή την αγορά, αντί να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή περιοχή σιδηροδρόμων, θα αρχίσουμε μια διαδικασία πολυδιάσπασης και δημιουργίας νέων εμποδίων. Και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε κόστος. Θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν όλους και ιδιαίτερα το Συμβούλιο να επιλέξει μια σωστή και δίκαιη λύση και για τα πολιτικά προβλήματα και για τα τεχνικά. Κυρία Γιάννα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς. Η επενδύση του κύριου Γιάνκερ έχουν σε στόχο ανάκαμψη και απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ένα προϋπολογισμό 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να δαπανηθούν. Με, τις ε, κρίσεις, με την κρίση τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια. Είσαστε έτοιμος να εξασφαλίσετε την απαραίτητη ευκαμψία ώστε αυτές οι επενδύσεις να μην καταλογίζονται στο, στο χρέος των κρατών μιλών και επίσης πώς θα αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη τα οποία εμποδίζουν τις διαμεθοριακές μεταφορές όπως γίνεται στη δική μου χώρα στα κεντρικά πυρηναία και για την απασχόληση. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα κοινωνικό πακέτο για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε τους ναυτικούς, έχουμε τους οδηγούς φορτηγών και έχουμε κοινωνικό dumping το οποίο θίγει πια και τους πιλότους των αεροπορικών εταιριών. Πώς Πότε θα μπορούμε να περιμένουμε από εσά, κύριε Επίτροπε, να παρουσιάσετε ένα πακέτο για το κοινωνικό ντάμπινγκ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τα δύο ερωτήματα. Το πακέτο επενδύσεων που αναφερθήκαμε προηγουμένως είχα πει ότι είναι μια σαφής ε, δέσμευση του Προέδρου της Κομισιόν ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να έρθουμε ενώπιόν σας μέσα σε τρεις μήνες για να σας προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το πακέτο 300 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις. Και εδώ εγώ είμαι απλώς ένας υποψήφιος επίτροπος αν πράγματι αναλάβω το, τα θέματα μεταφορών και διαστήματος είναι πολύ σαφές το κονδύλιο που θα πάει στις μεταφορές. Πιστεύω επίσης ότι σε αυτό το χώρο θα έχουμε σχέδια τα οποία θα είναι πολύ ελκυστικά για ιδιωτικούς επενδυτές σε εταιρική σχέση δημόσια, δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και επίσης θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε αυτά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να πράξει περισσότερα στον τομέα αυτό αλλά επίσης και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τα χρήματα μπορεί να προσελκυστούν και να επενδύσουν και αυτές για αυτά τα προγράμματα υποδομών. Τώρα, εάν πρόκειται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές. Το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει ήδη τροποποιηθεί και υπάρχουν ρήτρε ευκαμψίες που έχουν τροποποιήσει την αρχική μορφή αυτού του συμφώνου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις από τους δημόσιους πόρους και να εξακολουθήσουμε να έχουμε μία δυνατότητα χωρίς να θίξουμε το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την επερχόμενη Κομισιόν. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μοσκοβιτσί και ο κύριος Κατάινα καθώς και ο κύριος Δομπρόφσκης θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι ακόμα και στο τωρινό πλαίσιο τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα για τις μεταφορές θα μπορέσουν να προετοιμάσουν αυτό το πακέτο, την εφαρμογή αυτού του πακέτου επενδύσεων που ανέφερα. Ο Ζωσμπαχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε, υποψήφια επίτροπε. Οι ερωτήσεις μου αφορούν και εμένα τα δικαιώματα των επιβατών και χαιρετίζω τις δηλώσει και τις απαντήσεις που δώσατε στους προηγούμενους συναδέλφου για την διατροπικότητα και την επιβολή των δικαιωμάτων της ε, προστασίας του σεβασμού των δικαιωμάτων των επιβατών. Πολύ σωστά ξεκινήσατε. Θα ήθελα συγκεκριμένα να ρωτήσω εάν κατά την επεξεργασία των δικαιωμάτων των ε, επιβατών θα θέσετε τον ε, επιβάτη πάντα στο επίκεντρο της προσοχής, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Και επίσης υπάρχει μια σειρά ε, νομοθετημάτων, κυρίως για τις ενέργειες μεταφορές, συγκεκριμένα η οδηγία 261, Υπάρχουν διαφορές, αποκλίνουσες απόψεις ε, και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να αναλάβουν ένα κατά κάποιον τρόπο συνταγματικό ε, ρόλο, ένα νομοθετικό ρόλο θα έλεγα. Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το νομοθετικό έργο και έτσι το ζήτημα έμεινε στα χέρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να κρυθεί. Πώς μπορείτε λοιπόν νομίζετε να αντιμετωπίσετε αυτό το αδιέξοδο και να μας βγάλετε από τη το θέμα αυτό της 261 απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Συμφωνώ απολύτως ότι αν δεν είναι αρκετά σαφείς οι κανόνες, προφανώς αναγκαστικά ε, παρεμβαίνουν τα δικαστήρια με τις αποφάσεις τους. Οι πρόσφατες δε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης των κανόνων περί δικαιωμάτων ε, των επιβάτων, αλλά και η απόφαση σχετική με τη δεύτερη χειραποσκευή, όπως ονομάζεται, ε, έχουν μεγάλη σημασία και θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς στην νομοθεσία μας. Εάν προκύπτουν τέτοια ζητήματα δηλαδή θα πρέπει πάντοτε να διευκρινίζονται οι ε, διατάξει έτσι ώστε και να είναι σεβαστή η νομολογία και οι αποφάσεις του δικαστηρίου αλλά και όπως σωστά αναφέρεται να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής ο επιβάτης. Νομίζω ότι εάν δεν πιέζαμε τόσο για τα δικαιώματα των επιβατών θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα στις αεροπορικές μεταφορές. Θα είχαμε το overbooking, την ε, κράτηση δηλαδή πλεοναζουσών θεσεών που έχουμε ζήσει όλοι και φτάναμε στο αεροδρόμιο χωρίς να ξέρουμε αν θα μας βάλουμε μέσα στο αεροπλάνο ή όχι. Ε, ή θα είχαμε άλλου τύπου περιορισμούς που θα δυσκόλευαν πάρα πολύ τη ζωή μας, ιδιαίτερα για όσους ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους, με μικρά παιδιά. Αυτό λοιπόν και για να περάσω στο θέμα του Γιβραλτάρ, είναι λυπηρό, λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε να παγώσει μεγάλο κομμάτι αυτής της νομοθεσίας και βεβαίω η Επιτροπή έχει υποχρέωση τετερότητα ω προ την ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Ε, είμαι διτεθειμένο να συνεργαστώ με εσά και με το Συμβούλιο για να αναζητήσουμε έναν τρόπο να ε, λύσουμε το ζήτημα για να προχωρήσουμε στο νομοθέτημα. Η κυρία Κονσάλες Πένιας, αλλά και πάλι θα, θα παρακαλέσω τον υποψήφιο να τηρεί το χρόνο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η στρατηγική 2020 για την Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει μια περιεκτική και ευφυή και ανταγωνιστική ανάπτυξη. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση αναποτελεσματική των πόρων και επιβολή των συμφερόντων των επενδυτών στο σύνολο της κοινότητας. Και μέσα σε αυτά προκύπτει και όλο μικρότερη υποστήριξη για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυξάνονται οι αυτοκινητόδομοι, αυξάνονται τα αεροδρόμια τα οποία δεν έχουν κίνηση, ε, τρένα υψηλής ταχύτητος και δεν είναι όλα αυτά βιώσιμα όπως θα έπρεπε να είναι για την Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι οι πολιτικές μεταφορών θα χαραχθούν για τους λαούς της Ευρώπης, θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τους και θα λαμβάνουν υπόψη τη σημαντική, σημαντικό ρόλο που έχουν οι μεταφορές για την ευμάρεια και την κοινωνική συμμετοχή και δεν θα ακολουθούν μονάχα τα ιδιωτικά συμφέροντα ορισμένων μεγάλων φορέων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Θέτεται ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα έχει μονίμως μεγάλη σημασία στο μέλλον. Αυτό είναι οι δημόσιες μεταφορές. Είναι πολύ σαφές ότι ιδίως τους αστικούς ε, χώρους της πόλης της Ευρώπης δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις τωρινές συνθήκες μεταφορών. Όταν οι επιχειρήσεις μας και οι πολίτες μας χάνουν πάρα πολύ καιρό σε κυκλοφοριακές συμφορήσεις όπου καταστρέφουμε με την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου καταστρέφουμε το περιβάλλον μας και κάνουμε τις πόλεις μας χώρους που δεν είναι ευνοϊκοί για να ζει κανείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ε, αηφόρες δημόσιες μεταφορές γιατί αυτή θα είναι μια λύση που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και πιστεύω ότι και οι πολίτες, οι κάτοικοι των πόλεων θα την χαιρετήσουν και με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί και το θέμα αυτό το οποίο είναι τόσο σημαντικό στην Ευρώπη της απώλειας ενώ στα εκατό του ΑΕΠ μας γιατί τόσες πολλές ώρες κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μποτιλιαρίσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες των πολιτών, εγώ είμαι έτοιμο να προβούμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν προτάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση των μεταφορών και ξέρω ότι και με τις πόλεις είμαι έτοιμος να έρθω σε επαφή παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι τα κράτη-μέλη θα επικαλεστούν την επικουρικότητα και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το θέμα της προσβασιμότητας όταν δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς αγοράς όπως είναι η επιβολή δημοσίων υποχρέωσεων. Για Ευχαριστώ πολύ. Keith Taylor. Με, με, με τρομάξατε πρόεδρε, νόμιζα ότι δεν ήξερα ποιος είμαι. Κύριε Σεφκοβιτς, με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της δημόσιας υγεία στην πολιτική των μεταφορών, δεδομένου ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και αποδείξεις ότι προκαλείται καρκίνο αναπνευστικά νοσήματα, καρδιαγκιακά νοσήματα λόγω των ε, μεταφορών. Και θα ήθελα να συμφωνήσω ότι 26.000 θάνατοι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτα υψηλό νούμερο. Αλλά θα σας καλέσω και εγώ να θυμάστε ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 29.000 νεκρούς το χρόνο από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύτσοβιτς, για την ερώτησή σας νομίζω ότι αποδεικνύεται κατάφορα το πόσο οι μεταφορές είναι αλληλένδετες με τόσους άλλους τομείς πολιτικής και άρα έχουν κρίσιμη σημασία για την ευημερία του Ευρωπαίου πολίτη. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα, ρωτάτε, τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε κάθε δυνατή επιλογή ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι νεκροί από τροχέα στους δρόμους μας. Ήδη, όπως είπα, έχουμε αναλάβει μέτρα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο σημαντικά μέτρα, να βελτιώσουμε, να ξεχρονίσουμε τις υποδομές, το φωτισμό των δρόμων, να υποστηρίξουμε τις εξελίξεις αυτές όπου υπάρχει δυνατότητα και με, με ευρωπαϊκά ταμεία. Και πρέπει να δουλέψουμε σε καλύτερους, για καλύτερους στόχους αφορά τους σοφαρούς τραυματισμούς. 26.000 νεκροί είναι πολλοί, αλλά και οι 250.000 τραυματίες είναι πολλοί. Ο κύριος Τέιλορ. Ναι, για την, για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αναφέρθηκα μόλις τώρα στην απάντηση που έδωσα στη συνάδελφό σας η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Αν δούμε τι συμβαίνει στα αστικά κέντρα και κυρίως τις ώρες της κυκλοφοριακής αιχμής, είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ. Όπως είπα, πρέπει να φροντίσουμε να σεβαστούμε και τις πολύ λεπτές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο εισαρμοδέτες της Επιτροπής των κρατών μελών και των ε, τοπικών ή περιφερειακών αρχών, γιατί θα πρέπει να μπορούν οι, τα αστικά κέντρα να σχεδιάζουν μόνο τους τις μεταφορές όπως τις θέλουν για τον πολίτη του Εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ και με τις ε, ε, τοπικές περιφερειακές αρχές και με τις κρατικές αρχές, τις εθνικέ αρχές, για πλατφόρμες δημοσίων μεταφορών, για κινητικότητα καλύτερη, γιατί υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πόλεις μας εν γέννη. Ευχαριστώ κυρία Αιούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνο του 24% των εκπομπών καυσαερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδικές μεταφορές είναι το 18%. Παρ' όλα αυτά ε, τα οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικέ μορφές καυσίμων είναι ελάχιστα. Ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα όπως ε, οι κινητήρες με πεπιεσμένο αέρα ή οι ε, ηλεκτρικοί κινητήρες. Ή θα συνεχίσουμε να είμαστε όμοιροι των λόμπι των ορυκτών καυσίμων και να απαγορεύουμε σε αυτούς οι οποίοι να προχωρήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν νέες καινοτόμες μορφές κίνησης θα συνεχίσετε να είσαστε όμοιρος ε, των ε, πολιεθνικών εις βάρος των πολιτών ή θέλετε να κάνετε μία προσπάθεια για να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα υπέρ των εναλλακτικών. Μία δεύτερη ερώτηση. Η κυρία Ντελή είχε αναφερθεί στην γραμμή Τωρίνο Λιών και εσείς δεν αναφερθήκατε σε αυτό, την αγνοήσατε. Γνωρίζετε το ότι η γραμμή το Ρήνο ε, είναι μια παραδοσιακή σιδηροδρομική γραμμή και την χάνει ευρωπαϊκή βοήθεια σαν να ήταν υψηλής ταχύτητας, κάτι το οποίο είναι μια παράνομη χρήση των κοινοτικών πιστώσεων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τα εφή e, οχήματα, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ ε, να μην μείνουμε σε, στο, ε, παραδοσιακού τύπου διλήμματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι αδιέξοδα. Νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει, λέγουν ε, κάποιοι οι οποίοι προωθούν τις υποδομές ε, για τα καινοτόμα μέσα, ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τα FEE οχήματα, πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση του ηλεκτρισμού για την κίνηση, το υδρογόνο, τις κυψέλες υδρογόνου, πεπιεσμένου αέρα και οι νέες αυτές τεχνολογίες είναι σωστό να προωθηθούν αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα ΤΕΝ θα είναι σε θέση να καλυψεί και τις ανάγκες στις καινοτόμες αυτές μορφές κίνησης με εναλλακτικά καύσιμα. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι μπορούμε να δούμε περισσότερα εφή οχήματα στους δρόμους μας. Ο Γκέορκ Μάιερ. Ως ε, μη εγγεγραμμένος βουλευτής δυστυχώς βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να σας υποβάλω ερωτήσεις για επί λεπτά, αλλά μόνο για ένα λεπτό. Αλλά έχω να ρωτήσω το εξή. Ξέρετε ότι η Αυστρία είναι μετά την διεύρυνση προς Ανατολάς το είναι ένα κράτος ε, διέλευσης στις οδικές μεταφορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, τι έχετε να προτείνετε για, τις, ε, για τα σχέδια, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικά για την Αυστρία και αν, υπάρχει δυνατότητα για πραγματική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλα. Και μια πρόκειται για κράτος ε, διαμετακόμισης, ε, διέλευσης. Δεν θέλω να ρωτήσω αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα πολύ παλιά φορτηγά ε, που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τους πάντες. Τι θα κάνετε γι' αυτό λοιπόν. If I Εάν ε, μου επιτρέπετε η ερώτησή σας αφορά συγκεκριμένα την σύραγγα στην Αυστρία ή, ή Όχι, έχουμε δύο. Το COARM και το Σαν Μαρίν. Οι δύο αυτές σύραγγες με ενδιαφέρουν. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό πάλι σχετίζεται με, με τις προηγούμενες ερωτήσεις και το θέμα των ε, σειραγγών στους δρόμους. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση για τα TNT, για τα, για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα δηλαδή Μεταφορών. Επίσης γνωρίζετε ότι όλοι μας, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, συμφωνήσαμε ότι εφόσον θέλουμε αυτή η θετική μετακύληση να πραγματοποιηθεί με πραγματική αλλαγή στις υποδομές στην Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσουμε τα μέσα, τα κονδύλια που έχουμε στη θέσή μας σε πραγματικά έργα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στις υποδομές. Εξού και η επιλογή να ακολουθούν συμφωνημένα ε, έργα, μεθοδολογία, με διεξοδική συζήτηση που θα ε, ενέκρινε πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για μένα κάθε ένα από αυτά τα έργα είναι ισοδύναμο με νομοθεσία ευρωπαϊκή, γιατί το έχετε εγκρίνει εσείς. Πλέον έχει μείνει μόνο η εκτέλεση των έργων που έχετε ε, ψηφίσει και εγκρίνει. Έτσι θα χειριστώ για οδήποτε από αυτά τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων. Τώρα για να περάσω στο θέμα των ε, φορτηγών. Νομίζω ότι θα χρειαστώ περισσότερο από τα δευτερόλεπτα που μου λείπουν για τα πολύ μεγάλα φορτηγά, αλλά μια και ο πρόεδρος είναι τόσο ευστηρός με τον χρόνο θα πρέπει να περιμένω την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Κριστίν Ρεβόντα Αλόν, Μπονφουά. Ευχαριστώ πρόεδρε. J'ai bien compris votre détermination pour faire en Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το σιδηροδρομικό πακέτο να, να συζητηθεί στο σύνολό του. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει κίνδυνος ε, να μην καταλήξουμε κάπου. Θα εγκαταλείψετε σε αυτή την περίπτωση τις προσπάθειες για την τεχνική συμφωνία. Για τη συμφωνία στα τεχνικά θέματα πάνω στα οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και έχουν βρεθεί και κοινοί τόποι. Τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Σιδηροδρόμων, η οποία μειώθηκε ο προϋπολογισμός, οποίας μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά 5%. Αυτό πώς επηρεάζει το τεχνικό κομμάτι, πώς προβλέπετε εσείς να λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή με περισσότερες αρμοδιότητες και μικρότερο προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ κυρία σχετικά με τις εξωτερικές υπηρεσίες πράγματι μου ξανάρχονται αυτά από το παρελθόν. Ήμουν υπεύθυνο για τις ε, διαπραγματεύσεις των νέων αυτών ρυθμίσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Πάντως είναι σαφές ότι η υπηρεσία σιδρομική η ευρωπαϊκή είναι στην φάση οικοδόμησης, δημιουργίας και ολοκλήρωσης και είναι μια υπηρεσία για το μέλλον. Εγώ θα ανέμενα, αν θυμάμαι καλά, 43 επιπλέον θέσεις προσωπικού να δοθούν στην υπηρεσία αυτή, ε, που σε κάποια φάση θα αυξήσουν το προσωπικό τους γύρω στα 200 άτομα. Είναι σημαντική αύξηση αυτή. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό σε ένα ευρύτερο κλίμα μειώσεων 5% ε, στο σύνολο των εξωτερικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών. μπορούμε να το πετύχουμε μέσω της χρηματοδότησης ε, των νέων εμπειρογνωμόνων που οργάζονται για την συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω των ανταποδοτικών τελών. Ξέρετε ότι θα χρεώνουν για τις αδειοδοτικές τους ε, δραστηριότητες. Η υπηρεσία αυτή ε, είναι κάτι το οποίο αναμένεται ιδιαίτερος από την βιομηχανία της ηροδρομική θέλουν να, να απαλλαγούν από τις 26.000 εθνικούς κανόνες που εφαρμόζονται σήμερα και να μειώσουν και την, τον χρόνο αδειοδότησης νέων, νέου υλικού σιδηροδρομικού, τροχαίου υλικού και πρέπει να περνάει από εθνικές υπηρεσίες πολλαπλές ενώ τώρα τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα και η τεκμηρίωση θα είναι ταυτόσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, τα χρήματα που θα δαπανίσουν οι υπηρεσίες αυτές θα είναι χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν σωστά και έτσι θα καλύψουμε την αύξηση του προσωπικού. Και τώρα περνάμε στις ερωτήσεις από την Επιτροπή Ήτρε και καλωσορίζω τον πρόεδρό της, κύριο Μπούζεκ, η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε υποψήφι, επίτροπε, από τις μεταφορές πάμε στο διάστημα και έχω ερώτηση για το Γαλιλαίος. Είναι ένα από τα ε, μεγαλειώδη εγχειρήματα της Ευρώπης που έχει υποστηριχθεί ανέκαθεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον επιβεβαιωθείτε ε, στον τουρισμό αυτόν, θα συνεχίσετε με, την ίδια, ε, με τον ίδιο ενθουσιασμό στο έργο αυτό του Γαλιλαίου όπως και προκατοχό σας και επίσης για την ανάπτυξη του Γαλιλαίου έχετε πει ε, από την αρχή ότι σας ενδιαφέρει το θέμα των δορυφόρων, αλλά είχαμε προβλήματα στην ε, εκτόξευση των δύο τελευταίων δορυφόρων. Θα γίνει λοιπόν κάτι. Επίσης για το θέμα των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και τη πνευμηχανική τοκτησία στο Γαλλίο, γιατί ασφαλώ θα χρειάζεται κάποιο είδου αδειοδότηση για την πρόσβαση στα δεδομένα. Επίση, ε, η χρήση τόσο εμπορική όσο και από κρατικέ δημόσιε υπηρεσίε για το Γαλλίο. Θα με ενδιαφέρει να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιμπλερ για την πρώτη σας ερώτηση. Απερίφραστα ναι, διότι έχουμε εργαστεί για τόσα χρόνια με το ε, εγχείρημα αυτό του Γαλιλαίου. Ο προκάτοχος μου κύριος Σταγιάν ήταν αυτός ο οποίος τακτοποίησε τα του Γαλιλαίου. Έχουμε μια καλή ομάδα που δουλεύει για το έργο αυτό. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή νομίζω γιατί σήμερα έγινε ακόμη μια ε, έρευνα, ε, μια συνάντηση στην ε, Μόσχα, μια συζήτηση στη Μόσχα που ήθελε να διερευνήσει ακριβώς ποια ήταν τα προβλήματα, γιατί, γιατί εμφανίστηκε αυτό το injection anomaly, αυτό το πρόβλημα έγχυσης και πώς μπορούμε να σώσουμε τους δορυφόρους γιατί αν δεν μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε καλό θα είναι τουλάχιστον να μην τους χάσουμε τελείως ακόμα και βρεθούν σε διαφορετική τροχιά θα πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία τους στο διάστημα αλλά πάλι εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά αποτελέσματα από την έρευνα αυτή, από την Επιτροπή Έρευνας Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του, της θέσης σε τροχιά, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ε, ολίσθημα αυτό ε, ή, εν πάση περιπτώσει, για να είμαι και πιο σαφής, εγώ θα ήθελα να διαρευνηθούν διεξοδικά όλα τα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένω εμφανίζονται για να είμαστε σίγουροι ότι αναπτύσσεται σωστά το έργο. Ε, στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε την, το REN5 με τον τέταρτο δορυφόρο και άρα θα μπορεί το έργο Γαλιλαίος να αναπτυχθεί σε, αυτό το στερέωμα που ονομάζεται Daily Service. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς, σας χαιρετίζω και σας καλωσορίζω για την παρουσία σας. Καταρχήν, είχα την ευκαιρία να δω το έργο σας στην τωρινή θητεία της Κομισιόν Δείξατε ενεργητικότητα και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Σας εύχομαι να συνεχίσετε και στην επόμενη Επιτροπή. Είδα να έχετε ένα σαφές όραμα σε σχέση με την ανάπτυξη των θεμάτων στο χαρτοφυλακιό σας που είναι εκτενές και πολύπλοκο, έχει πολλές δυνατότητες. Θα ήθελα όμως να σας θέσω ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένο. Ποια είναι η άποψή σας για την διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες είναι οι κέρδιες πρωτοβουλίες που έχετε σαν στόχο να ξεκινήσετε έχετε την πρόθεση να παρουσιάσετε μια πολιτική για εκτοξευτές ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να είναι από τα κυριότερα προβλήματα που θα συζητηθούν το Δεκέμβριο στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ. Ποια άλλα μέτρα επίσης θα λάβετε στον τομέα της εξερεύνησης του διαστήματος που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ <clears throat> για τα θερμά σας λόγια, αλλά νομίζω ότι η ενεργητικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι κέρια στοιχεία για την διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα θέματα μεταφορών ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και για τη διαστημική μας πολιτική. Έχουμε μπροστά μας, τα έλεγα, τα πιο κέρια πέντε χρόνια για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική πιο σημαντικά από ό,τι ποτέ. Θέλουμε ο Γαλιλαίος να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του. Δηλαδή σχεδόν 30 δορυφόρους, εξαρτάται πόσοι από αυτούς θα είναι σε τροχιά και ποιοι, πόσοι θα είναι σαν δορυφόροι ε, ενδεχόμενης αντικατάστασης. Επίσης θέλουμε να πράξουμε το ίδιο και με το πρόγραμμα Κοπέρνικος, όπου θέλουμε να αναπτύξουμε 12 δορυφόρους παρακολούθησης της γης, γιατί ο Γαλιλαίος είναι περισσότερο για το σύστημα ε, εντοπισμού και επίσης και για την ε, διατήρηση της ακρίβειας των ατομικών ρολογιών, ώστε παραγωγικά να γίνεται σαφής η χρονική στιγμή των ε, συναλλαγών που γίνονται σε χρηματοπιστωτικά ανταλλακτήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρώπη να εξασφαλίσει την ε, ανεξαρτησία της και όχι να βγει από το παιχνίδι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε την αυτόνομη πολιτική διαστήματός μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους εκτοξευτές υπάρχουν ε, αναλύσεις που έχουν γίνει και προπαρασκευαστική εργασία για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε την Αριάν 5 ή την Αριάν 6 και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μονάχα ένα μεγάλο εκτοξευτή όπως είναι η Αριάν 5 και ένα μικρό εκτοξευτή όπως είναι το Ρέγκαν, αλλά και κάποιον ενδιάμεσο για τις ε, ε, εκτοξεύσεις που γίνονται από ξένους πυράβλους αυτή τη στιγμή. Λουτουλόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η υποψηφία επίτροπε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα για να σας ρωτήσω για την πολιτική του διαστήματος που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης ε, που θα αναπτυχθεί με το έργο Καλλιλέως. Πιστεύετε ότι μπορούν να υπάρχουν συνεργατικές σχέσεις και να αναλάβει με τον τρόπο αυτόν η νέα υπηρεσία νέα καθήκοντα όπως με το Κοπέρνικος αλλά και με αντίστοιχα ε, έργα τα οποία από μόνα τους θα μπορούσαν να φανούν είτε πολύ δαπανηρά είτε και περιτά. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που μπορώ να σας απαντήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα τώρα γιατί ξέρω ότι θα με καταλάβετε αν μιλάω σλοβακικά. Για το μέλλον λοιπόν και την ε, υπηρεσία αυτή της πράγας. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε εδώ αναπτύξει προτεραιότητες για το μέλλον με την ε, υπηρεσία αυτή και το γεγονός ε, ότι ξεκινάει αυτή η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και εμπορικά ο Γαλιλαίος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το έργο αυτό για τον Ευρωπαίο πολίτη αλλά και για την ε, επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ε, ευρύτατα καθήκοντα να επιτελέσει. Εδώ μιλήσαμε για το Κοπέρνικο νωρίτερα. Πάνω από 100 αεροδρόμια της Ευρώπης αξιοποιούν το σύστημα αυτό διότι είναι πολύ πιο φθηνή η τεχνολογία αυτή και πολύ πιο σύγχρονη. Επίσης είμαι πεπισμένος ότι η χρήση και αξιορολόγηση, αξιοποίηση ε, στοιχείων που μπορούμε να αντλήσουμε από το σύστημα Κοπέρνικος θα πρέπει να ε, γίνει κατά τρόπον ώστε οι πληροφορίες να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Με την προετοιμασία που έκανα για τη σημερινή ακρόαση διαπιστώνω ότι τα δεδομένα του Κοπέρνικου σημαίνουν πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά ε, στην, για να είμαι ακριβής σημαίνουν νούμερα της τάξης του 1 στην ε, του 1 με 15 μηδενικά, γιατί δεν μπορώ να σας διαβάσω το νούμερο, ε, και άρα τα δεδομένα αυτά σημαίνουν τεράστιες δυνατότητες και για την Επιτροπή, πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν, πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Frontex ή κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως η περιβαλλοντική, η υπηρεσία, η υπηρεσία για την ασφάλεια στις τεράστιες μεταφορές. Δηλαδή έχει τεράστιο δυναμικό για εφαρμογές. Ευχαριστώ ο κύριος Κρικέ, ο οποίος κάθεται και πίσω σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφι Επίτροπε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το διάστημα, μια και είναι η σειρά του, αλλά και ως Αντιπρόεδρος Επιτροπής των Μεταφορών για τις μεταφορές. Για το διάστημα Υπάρχει μια πρόταση για υποστήριξη βιομηχανική των χερσαίων εφαρμογών του Γαλιλαίου. Αυτό έχει γίνει με την προηγούμενη Επιτροπή. Αυτό υπάρχει σε επίπεδο, σε στάδιο προετοιμασίας και αφορά ύψος αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και δεύτερον σκοπεύετε να υποστηρίξετε περισσότερο τις δυνατότητες εκτόξευσης και κυρίως βαρέως βελνε, βαρέως ε, επίπεδου. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ε, για τις οδικές μεταφορές και για τις μεταφορές γενικότερα και τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους που έπρεπε να λάβετε κάποια μέτρα. Για τις οδικές μεταφορές έχετε κάτι επιπλέον να μας πείτε για την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο του Γαλιλαίου στο βαθμό που μπορούμε και όπου μπορούμε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ώστε να υπάρξουν νέε αποδέκτες για το σύστημα και να είναι ε, συμβατά τα συστήματα όπως το οίκο παραδείγματι με το Γαλιλαίο. Σε όλος ο εξοπλισμός ο οποίος σχετίζεται με την έρευνα και διάσωση στις διάφορες, τις διάφορες περιοχές κρίσης, όπου έχουμε σαφέστατες ρυθμιστικές εξουσίες, μπορούμε να επιβάλλουμε, να είναι συμβατός ο εξοπλισμός με το Γαλιλαίο. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε στενά σε συνεργασία και με τον κλάδο και με τις υπηρεσίες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν ε, αρχίσει να εκπέμπει σήμα ο θα έχει ε, μαζική αποδοχή και θα φέρει τους καρπούς του απευθείας στον, ε, στην οικονομία της Ευρώπης, στις επιχειρήσεις της Ευρώπης, γιατί θα είναι πολύ πιο ακριβής ο Γαλιλαίος θα έχει δίνει δηλαδή πολύ πιο ακριβή στοιχεία αναγνωρίσιμα από ό,τι γνωρίσουμε τώρα από το σύστημα GPS και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας. Ε, λαμβάνονται όμως και όλα τα μέτρα, αναλαμβάνονται όμως και όλα τα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του Γαλιλαίου. Για τους εκτοξευτές ε, είναι μεγάλου βεληνικού έργου, έργο, αλλά βεβαίως ε, τάσσομαι υπέρ ιασδήποτε επιλογής που θα μας εξασφάλιζε αυτονομία στο διάστημα. Ευχαριστώ επόμενο μιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να δώσω τη δυνατότητα στον κύριο υποψήφιο επίτροπο να μιλήσει σλοβάκικα και γι' αυτό θα θέσω ερώτημα στα τσεχικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να αναφερθεί ο κύριος Επίτροπος για τα θέματα θαλασσίων μεταφορών και εσωτερικών υδατίνων δρόμων ε, που χρησιμοποιούνται μόνο σε περιορισμένο επίπεδο 15% σε ορισμένε περιπτώσει. Τι θα κάνετε λοιπόν για άλλους ποταμούς, τι θέλετε να κάνετε. Στην Λευκορωσία θέλουν να συνθέσουν τον Δυτικό Δβίνα στον Δνήπερο κάτι το οποίο θα επιταχύνει τις ε, διελεύσεις κατά τέσσερις φορές από τη Μεσόγειο στην Βαλτική θάλασσα. Θα ήθελα να ξέρω αν θέλετε να υποστηρίξετε το φιλόδοξο σχέδιο του πρόεδρου μας, του Μίλο Ζέμαν, σύνδεσης μεταξύ ε, Δούναβη και Όντερ και Έλβα. Με τη σύνδεση λοιπόν αυτή θα, έχουμε, θα, θα υπάρχει σύνδεση τριών ευρωπαϊκών ε, θαλασσών, αλλά με τον τρόπο αυτό θα παραβιαστεί και η γερμανική νομοθεσία γιατί το Βραδεμβούργο και η Σαξονία έχουν ήδη βγάλει ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο ε, Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα και να σας ευχαριστήσω για το ερώτημά σας. που δείχνει και πάλι τη σημασία του να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό το οποίο υπάρχει στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Οι δυνατότητες λοιπόν οι οποίες υπάρχουν σε αυτό το τομέα είναι φυσικά περιορισμένες λόγω του προϋπολογισμού μας αλλά χαίρομαι και για την υποστήριξη που έχω λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε το ίδιο επίπεδο πόρων όπως και στην προηγούμενη θητεία, στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο μάλλον, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε σχέδια για εσωτερικές διαδρομές στον Δούναβη, μπορεί να ανανεωθεί ο στόλος των ποταμοπλοίων, γιατί υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. <clears throat> μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε τις λιμανικές υποδομές και των, ε, τις υποδομές των καναλιών στις παραδουνάβιες περιοχές. Μας ενδιαφέρει όμως να προχωρήσουμε και σε καλύτερη κατάρτιση του, των εργαζομένων στις εσωτερικές υδάτινες διαδρομές. Πολλές φορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Για τα σχέδια που ανέφερε ο κύριος βουλευτής, το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι είναι συμβατά με τα τέντη και με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουμε στον τομέα αυτό. Ο κύριος Κόμπορν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα συμφωνούσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως στον τομέα μεταφορών δεν θα πρέπει να κατασπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων σε προγράμματα υψηλού κύρους που δεν ευνοούν και δεν ωφελούν κανένα από τους ε, φορολογούμενους. και το τελευταίο τέτοιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Νότια Ευρώπη. Συμφωνείτε ότι αυτά τα σχέδια μεταφορών είναι και αυτά ένα είδος φαντασιώσεως που έχει σαν στόχο να μιμηθούμε τους Αμερικανούς. Το πρόγραμμα Γαλιλαίος και Κοπάνικος δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και των Βρετανών υπηκόων. Το να μπορεί κανείς να εξασφαλίζει ότι μπορεί να φορολογεί όλα τα αυτοκίνητα των Ευρωπαίων όταν κινούνται στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος, ενώ υπάρχει μια λιτότητα που καλύπτει όλους. Θα χρησιμοποιήσετε τη θέση σας να σταματήσετε αυτό το παράλογο, το μεγαλόσχημο σχέδιο το οποίο είναι σε βάρος των φορολογουμένων. Σίγουρα η ιδιωτική αγορά είναι σε πιο καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διαστημικής βιομηχανίας από ό,τι κράτη ή η νομενκλατούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως υποψήφιος επίτροπος θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και για αυτό το ερώτημα. Κατανοώ βέβαια ότι εδώ φαίνουμε απόψεις που θα έπρεπε να περιληφθούν στη συζήτηση. Πιστεύω όμως και από την προηγούμενη δήλωσή μου θα έχετε κατανοήσει ότι δεν συμμερίζομαι με, με τις απόψεις που έχετε εκφράσει για την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος και φυσικά δεν συμφωνώ και με την περιγραφή που έχετε δώσει για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα αυτό. Γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα διαστημικό πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία μας στον τομέα αυτό και την αυτονομία μας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διάστημα και δεν είναι μονάχα θέμα κύρους, μονάχα και ακτινοβολίας, δεν είναι θέμα κύρους, δεν είναι θέμα ακτινοβολίας. Το χρειαζόμαστε για την τεχνολογία μας ε, εχμής, για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα συμφόρησης της πόλης μας. Τα χρειαζόμαστε και για τον τραπεζικό μας τομέα ακόμα. Αν ρωτήσετε τους συναδέλφους σας στο City του Λονδίνου, θα σας πούν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η σφραγίδα των ατομικών ορολογίων για όλες τις συναλλαγές που γίνονται στο City του Λονδίνου. Δεν θα πρέπει εδώ να εξαρτιόμαστε μονάχα σε ένα σύστημα όσο καλό και να είναι. Εμείς συνεργαζόμαστε φυσικά με το GPS, αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι αρκετά όρημη, αρκετά ανεπτυγμένη για να έχει τα δικά της συστήματα τα οποία από ό,τι γνωρίζω υποστηρίζονται και από τους Αμερικανούς εταίρους μας. Ευχαριστώ. Jetzt έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Όχι, ε, θέλω να επισημάνω ότι πάλι εδώ έχουμε τις ερωτήσεις Επιτροπή Σίτρε και θέλω να ευχαριστώ τον Πρόεδρο και δίνω το λόγο στην ε, κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ενιαίο οικονομικό και νοσηματικό χώρο απαιτεί και ενιαίο χώρο των μεταφορών. Ωστόσο, στην χρονική στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 23 διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το, η συζήτηση για την επιβολή διοδίων στους γερμανικούς δρόμους ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν ελοποιηθούν τα σχέδια της Γερμανίας, λαϊκιστές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης θα, χρειαστεί, θα θελήσουν να εφαρμόσουν αντίστοιχα συστήματα, πράγμα το οποίο οδηγεί σε δυσφορία, σε αισθήματα ε, δυσάρεστα και βέβαια οδηγεί και στον κατακαιρματισμό των μεταφορών και στον παραλογισμό τελικά. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο χώρο των μεταφορών. Δεν είναι δυνατόν τα εθνικά κράτη να κάνουν διακρίσεις ε, και αυτό να γίνεται ανεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν πώς στάσεστε σε περίπτωση επιβολής ενός ε, συστήματος επιβολής διοδίων κατά τρόπο ε, που επιβάλλει διακρίσεις. Σκοπεύετε να αναλάβετε δράση σε μελλοντική συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας. Ο πρόεδρος, νομίζω ότι πάλι και εσεί θα πρέπει να δώσετε μόνο σα την απάντηση για να αφήσετε χρόνο στον ερωτώμενο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε και κάποια προβλήματα. Έχουμε... Είμαστε καλοί στη δημιουργία υποδομών, αλλά δεν είμαστε πολύ καλοί στην συντήρησή τους επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα για δημιουργία υποδομών αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα προσέλκυσης ε, επενδύσεων για τη συντήρηση των υποδομών αυτών. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, ε, το τι θα γίνει με τα εξωτερικά κόστη και πόσο μπορεί να καλυφθούν αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοί να βρούμε πηγές χρηματοδότησης οι οποίες ε, να καλύπτονται και φυσικά από τους χρήστες των υποδομών σε σχέση με την ποσότητα βέβαια ε, και το ποσοστό χρήσης τους. Όταν διασχίζει κανείς την Ευρώπη με αυτοκίνητο και πληρώνει διόδια και στο τέλος ε, βλέπει κανείς ότι δεν ε, μπορεί να διακρίνει πολύ εύκολα προς τα έξω γιατί το παμπρίζ του έχει καλυφθεί από όλες τις βινιέτες που πληρώνει ε, υποχρεωτικά στις χώρες τις οποίες διασχίζει. Λοιπόν, το σύστημα θα πρέπει να γίνει πιο δίκαιο, ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρόνο χρήσης των υποδομών. Υπάρχει δυνατότητα η τεχνολογική και φυσικά η αρχή της έλλειψης διακρίσεων ε, είναι στη συνθήκη, είναι μια αρχή την οποία σέβομαι και θα σέβομαι. Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε ένα νέο μέσο, τον μηχανισμό για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, που θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα στους σιδηροδρόμους και στις οδικές μεταφορές. Στη χώρα μου επιμένουμε κυρίως στις δεύτερες. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και των δύο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τα προγραμματικά ομόλογα, τα project bonds, για να χρηματοδοτήσουμε επίσης και τους μηχανισμούς διασύνδεσης στην Ευρώπη. Ε, μία άλλη ερώτηση. Θα πρέπει να υπάρξει ένας επίτροπος ο οποίος στην ουσία να καταστεί αυτό που θα ονόμαζα ένας υπουργός μεταφορών, όχι μόνο κάποιος που θα σχεδιάζει. Έχουμε τα προβλήματα με το ρωσικό εμπάργκο, αυτό δεν θίγει μόνο ε, τους παραγωγούς οποροκυπευτικών και γαλακτοκομικών αλλά και τους μεταφορείς οι οποίοι μετέφεραν ακριβώς αυτά τα προϊόντα. Ε, θα ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Όταν αναφερθείτε στα, στα θέματα των σχέσεων με την Ρωσία θα παίξετε τον ρόλο του Υπουργού Μεταφορών Είδαμε επίσης το τι κάνει η Γαλλία σε σχέση με το χρόνο ανάπαυσης ε, των οδηγών φορτηγών. Ε, νομίζω ότι είναι κάποιες ιδέες οι οποίες ε, θα άρεσαν και σε μένα και σε σας. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Σεύκοβιτς, για την διασφάλιση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα διάφορα TNT. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει και στο Κοινοβούλιο για το ποια θα είναι η μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσουμε και τι κατανομή θα υπάρξει στον τομέα της χρηματοδότησης. Ένα ποσοστό δηλαδή της κάλυψης ε, της χρηματοδότησης ε, του Connecting Europe θα αφορά τις περιοχές οι οποίες υπάρχουν προβλήματα για το πέρασμα από τη μια χώρα στην άλλη και γενικά θα ασχοληθεί με τις αιστείες των προβλημάτων των ευρωπαϊκών μεταφορών. Ε, στην περίπτωση τώρα των προγραμματικών ομολόγων, νομίζω ότι σαν μέλος της Επιτροπής Μπαρόζο 2 εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ένα καλύτερο τρόπο χρήσης τους και να προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλους καινοτόμους τρόπους προσέλκυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στις ε, υποδομές και στην ανάπτυξη των υποδομών. Σε σχέση με το ρωσικό εμπάργο, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια του νέου συνόλου των επιτρόπων και θα προσπαθήσω να εκφραστώ πάνω σε αυτό και στις επαφές που θα έχουμε με τους Ρώσους εταίρους. Πείς μικρόφωνο επόμενος. Äh, elnök úr, äh, tisztelt Sefcsovics úr, az egyike a 9 äh, TNT folyosónak a... Ένα από τα εννέα ένας από τους νέους, από τους εννέα διαδρόμους των Τεντή είναι αυτός που συνδέει το Ρήνο με τον Δούναβη και θα είναι μια από τις σημαντικότερες συνδέσεις ανατολικά από τα ανατολικά προς τα δυτικά στην κεντρική Ευρώπη, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον ε, Ρήνο. Αυτό είναι τμήμα μια στρατηγική για το δούναβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σαν στόχο να προωθήσει την κινητικότητα και διατροπικότητα στου εσωτερικού υδάτινου δρόμου. Αλλά η ευρωπαϊκή δρόμη δεν είναι μονάχα σημαντική για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τα συνδυόμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη όπως είναι η Σερβία, η Βοσνία Ζεγοβίνα, η Μολδαβία, η Ουκρανία. Με ποιο τρόπο έχετε την πρόθεση να εξασφαλίσετε υποψήφιε επίτροπε ότι αυτές οι μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες θα έχουν και αυτές την χρηματοδοτική ικανότητα να εφαρμόσουν σχέδια τα οποία είναι κέρια και αυτά για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υδάτινων δρόμων. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Έχετε μεγάλο δίκιο ότι ο διάδρομος Ρήνου Δούναβη θα είναι πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ επίσης και για το ενδιαφέρον σας σε σχέση με χώρες όπως η Σερβία, η Μολδαβία, η Βοσνία Ζεγοβίνη. Πρέπει να πω ότι ενθαρρύνθηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι οι χώρες αυτές ενδιαφέρονται και έχουν ενθουσιασμό για τη στρατηγική του δύναμη. Ήταν μια από τις πρώτες μακροστρατηγικές που αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή του Δούναβη και νομίζω ότι η ελκυστικότητα αυτής της στρατηγικής είναι ότι χάρη στην συνολική αντιμετώπιση που είχε η Κομισιόν που καλύπτει κράτη-μέλη και γειτονικά κράτη μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων χρηματοδότησης και των ταμείων για να έχουμε σχέδια τα οποία είναι πιο ολοκληρωμένα με καλύτερη σύνδεση και μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι μια προσέγγιση λοιπόν που εγώ θα ήθελα να την υποστηρίξω ιδιαίτερα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η πρώτη μας προτεραιότητα και η κύρια εστίασή μας είναι να επιτύχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά και εν καιρό να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου για υδάτινους δρόμους. Ξέρουμε όμως ότι αυτοί οι δρόμοι δεν σταματάνε στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση τους και σε γειτονικέ χώρες. Αυτό θα είναι και ευνοϊκό για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί έτσι μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση, την εμπειρία, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Είναι καλό για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Η δίκη Μέιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις συγκεκριμένες νομίζω ερωτήσεις. Πρώτον, ε, για το φιάσκο του προηγούμενου μήνα. Εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή Θα ήθελα να μάθω όμως ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες από την αποτυχία της, ε, της θέσης έτροχιά των δύο ε, δορυφόρων και τι θα κοστίσει στους φορολογούμενους. Δεύτερον, με ποιο τρόπο θα μειώσετε την γραφειοκρατία στον τομέα των μεταφορών. Και τρίτον, κύριε υποψήφιε επίτροπε, τι θα κάνετε με τις κίτρινες κάρτες των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας σχετικά με τις εκτοξεύσεις Ε, ε, τον Αύγουστο για τον Γαλιλαίο. Είναι ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Και τα θέματα αυτά και οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Εμείς απογοητευθήκαμε ιδιαίτερως βέβαια για το συμβάν. Ε, κάποιες, κάποια πρώτα συμπεράσματα από το άτυχο αυτό συμβάν δείχνουν ότι οι δορυφόροι μας είναι μεν καλοί, είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι και λειτουργούν πάρα πολύ σωστά. Και η δυσλειτουργία προκλήθηκε από το τελευταίο τμήμα του πυράβλου, του εκτοξευτήρα. Και γίνεται μια συνεχής τεχνική έρευνα για το πώς συνέβη το ατύχημα αυτό και πώς θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Είμαστε σαφείς σε αυτό. Δεν μπορούμε εμείς ε, να, να συνεχίσουμε με αυτού του είδους ε, τους εκτοξευτές διότι ε, θα πρέπει τα χρήματα και τα χρήματα των φορολογουμένων να μην χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχουμε μια ειδική σύμβαση για τα επόμενα δύο χρόνια για τρεις εκτοξεύσεις. Μπορεί να μεταφέρει ο εκτοξευτήρας αυτός με τον οποίο έχουμε συμφωνία ε, τέσσερις δορυφόρους και όχι δύο είναι ευρωπαϊκής ε, σχεδίασης και νομίζω ότι με τους Αριάν, τις εκτοξεύσεις Αριάν θα μπορέσουμε εν πολύς να αντισταθμίσουμε τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τις εκτοξεύσεις αέρους. Τώρα για την γραφειοκρατία. Ε, φυσικά και θα είμαστε απολύτως σοβαροί στην αντιμετώπιση της. Θα χρησιμοποιήσουμε και τα REFIT για να αξιολογήσουμε τις νομοθεσίες οι οποίες θα χρήζουν τροπολόγησης και αλλαγής. Και εφόσον έχετε συγκεκριμένες ιδέες για το ποιες ε, ε, νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να καλυφθούν εδώ, θα συνεργαστώ μαζί σας όσο στενότερα μπορώ, σεβόμενοι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο κύριος σας ευχαριστώ. Είμαι εδώ στο βάθος κύριε Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα. Θα αναφερθώ στις γραπτές σας απαντήσεις για την αηφορία στις μεταφορές. Είναι απογοητευτικές λίγο γιατί δεν είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό θα σας βοηθήσω να γίνετε πιο συγκεκριμένους. Λοιπόν θα δούμε πώς θα τα πάτε. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, ότι στα πλαίσια του πακέτου και των στόχων 2030 δεν υπάρχουν και πάρα πολλά για τις μεταφορές, ενώ η Λευκή Βίβλο ε, φαίνεται ότι θα χρειαζόμαστε για τις μεταφορές συγκεκριμένα ε, μέσα για μετά το 2020, ε, τι θα γίνει με τις οδηγίες οι οποίες θα εκκρεμούν μετά το 2020 τώρα για τις αερομεταφορές. Η ΚΑΟ θα πρέπει να δώσει προτάσεις για τις παγκόσμιες αερομεταφορές το 2016. Θα πιέσετε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί αν αφήσετε το ΙΚΑΟ μόνο του, τότε δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να γίνω πιο συγκεκριμένος στις αξιολογήσεις μου. Και σας ευχαριστώ και για τις ιδέες τις οποίες προτείνατε. Σχετικά τώρα με την κατάσταση μετά το 2020 και σε σχέση με τους στόχους σαν παράδειγμα για τα βιοκαύσιμα. Είστε εμπειρογνώμων σε σχέση με αυτά και γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα με τη χρήση των, ε, πρώτης, των ε, βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα λοιπόν ε, με τα εναλλακτικά καύσιμα. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες και οι οποίες ελπίζω ότι μετά το 2020 θα βοηθήσουν. Ε, και σε σχέση με τους στόχους της μόλυνσης ε, της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα στις πόλεις μας, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, οι νέες τεχνολογίες και οι νέες μορφές μεταφορών που να είναι καθαρές, που να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες τεχνολογίες είναι απαραίτητες και θα πρέπει να είναι και σωστά διατροπικές με την έννοια ότι θα δώσουν κίνητρα στους ε, πολίτες να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην κατοικία τους. Αυτό θα μειώσει τη μείωση της ατμόσφαιρας ε, και θα απελευθερώσει τους δρόμους. Ε, Αυτό είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα απαντήσω στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας. Τώρα, για το ΙΚΑΟ. Ξέρετε ότι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο λίγων περίπλοκη, διότι δεν είμαστε μέλη του ΙΚΑΟ αλλά παρατηρητές. Επαφιέμεθα δηλαδή στην συνεργασία με τα κράτη-μέλη και στο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΙΚΑΟ. Θα χρησιμοποιήσω όλες τις επαφές τις οποίες έχω στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών με τους υπουργούς που θα είμαι σε επαφή έτσι ώστε οι θέσεις ε, του Συμβουλίου να είναι σωστά συντονισμένες. Ένα ερώτημα για τις οδικές μεταφορές και τον ανταγωνισμό στις οδικές μεταφορές. Είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτή <clears throat> να υπάρξει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και αυτό δεν θα πρέπει να μείνει μονάχα στα χέρια των κρατών μελών. Είδαμε τους τελευταίους μήνες πολλά προβλήματα και ιδίως σε ό,τι αφορά την ε, διαρρύθμιση για το χρόνο ανάπαυσης και χρόνο οδήγησης. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, δεν θα θεωρεί ότι η ανάπαυση στην καμπίνα του φορτηγού είναι πραγματικός χρόνος ανάπαυσης και κινδυνεύουν οι οδηγοί με πρόστιμα 3.000 ε, ευρώ. Ενώ σε άλλες χώρες επιτρέπεται η ανάπαυση στην καμπίνα του φωτιγού. Εσείς ως Επίτροπος τι δράση θα αναλάβετε για να αντιμετωπίσετε τα θέματα της εφαρμογής νομοθεσίας αυτού του είδους ώστε να εφαρμόζεται με ισόρροπο τρόπο σε όλες τις χώρες και ακολουθώντας αυτό που είπε ο κύριος Ρικέ, τι θα κάνετε με τη φιλελευθερωποίηση σε επίπεδο καμποτάζου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Πιστεύω ότι όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτεται καταδεικνύουν αυτό το οποίο είπα ήδη και εγώ, ότι αυτό που είναι απαραίτητο στις οδικές μεταφορές είναι να υπάρχει μια σε βάθος εξέταση της τωρινής κατάστασης του μεταφορικού τομέα και τις τωρινές κατάστασεις της νομοθεσίας και θα πρέπει να κάνουμε τα εξή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε την νομοθεσία αυτή, δεύτερον να την απλοποιήσουμε και τρίτον να εμπλέξουμε τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν τα πράγματα και θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους ώστε να εξασφαλίσουμε <clears throat> ότι θα μπορέσει να υπάρξει σεβασμός των κοινωνικών τους δικαιωμάτων στον τομέα των μεταφορών και θα έχουν μια κοινή πλατφόρμα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και φυσικά ό,τι προκύψει από όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η πρακτική αυτή που αναφέρατε για τη Γαλλία για τον χρόνο ανάπαυσης ε, μπορώ να σας πω ότι το ίδιο ισχύει και στο Βέλιο. Δεν έχω δει σε άλλες εθνικές νομοθεσίες μια τέτοια σαφή μορφή περιορισμού ότι δεν μπορεί κανείς να περάσει το χρόνο ανάπαυσης μέσα στην καμπίνα του φωτιού. Προτού όμως καταλήξουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα και που θέλω να συνεχιστεί, είναι να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέσω του λεγόμενου πιλότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συστήματος αυτού που μας επιτρέπει να λύσουμε προβλήματα όταν δεν υπάρχει επακριβής εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέσουμε το θέμα αυτό με τις αρχές του Βελγίου και της Γαλλίας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική λύση η οποία δεν θα είναι διακριτικού χαρακτήρα και θα σέβεται την τωρινή κείμενη νομοθεσία. Κόσμος Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχω την εξή ερώτηση. Για την κατασκευή δρόμων. Στη χώρα μου έχουν κατασκευαστεί πολλοί δρόμοι. Αλλά με κάποιο παράδοξο τρόπο, δηλαδή γίνονταν διάφορα κομμάτια αυτοκινητοδρόμων χωρίς όμως σύνδεση μεταξύ τους. Κάπου ξαφνικά σταμάταγε ο δρόμος. έργο υποδομών πρέπει να είναι έργο το οποίο παραδίδει αποτέλεσμα 100% λειτουργικό. Λοιπόν, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται οι δρόμοι. Να μην γίνεται τμηματικά η κατασκευή. Έτσι ώστε αν δεν είναι ε, ολοκληρωμένος ο δρόμος να μην μπορεί να παραδίδεται. Θα πρέπει να συνδέεται το ένα σημείο, το ένα σημείο Α με ένα σημείο Β. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Πολωνία. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε αρκετά Δεν πιστεύω ότι ήταν εσκεμμένες πάντοτε αυτές οι επιλογές. Μερικές φορές έχουν να κάνουν με την ε, διαδικασία των προμηθειών και ενστάσεις που μπορούν να τραβήξουν επιμακρών ε, η ανάγκη για την εξαγωγή μιας πολύ αυστηρής περιβαλλοντικής μελέτης για το συγκεκριμένο έργο. Πάντως συμφωνώ μέσα ότι θα πρέπει ε, ιδιαίτερα στο πώς θα κριθεί ένα έργο, δηλαδή το να παραδίδεται ένα έργο το οποίο ε, είναι ε, χρηστικό, ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Δεν μπορεί να πηγαίνει δηλαδή κάποιος σε ένα δρόμο και ξαφνικά να τελειώνει ο δρόμος και να μην μπορεί να συνεχίσει με τις ίδιες συνθήκες μεταφοράς την πορεία του, να αλλάζουν δηλαδή οι συνθήκες μεταφοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε πολλές συμφορήσεις και πολλά άλλα προβλήματα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Και είναι προφανώς πολύ πιο σημαντικό να εστιμαστούμε στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και βελτιώνουν τις υποδομές σε ολόκληρο το χώρο, έργα τα οποία θα γίνεται κατανοητό και για τον Ευρωπαίο πολίτη ότι βελτιώνουν την κατάσταση στην περιοχή του. Που θα μπορεί να δει ότι έχει καλύτερες μεταφορές στην πόλη του ή στην περιφέρεια του. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και με τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Πολιτικής, ε, με την DG Move για την πολιτική των μεταφορών της κινητικότητας. Ευχαριστώ πολύ, Ιζαμπέλα Ντεμόντα. Θα ήθελα να επανέλθω στο του καμποτάζ. Εσείς είπατε στην εισαγωγή σας ότι είναι ένα σύστημα χρήσιμο έτσι ώστε να μπορούν να μην κυκλοφορούν κενά ε, τα μεγάλα φορτηγά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει διορθωθεί από τις ε, οδηγίες οι οποίες ισχύουν και οι οποίες δημιούργησαν ψευδεστήσεις. Αναφερθήκατε και στα θέματα των καινοτομιών. Οι καινοτομίες σε τέτοια φαινόμενα μπορούν να είναι χρήσιμες. Thank Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ πράγματι ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας πήρε μέρος ε, σε μια συνάντηση όπου τέθηκε το θέμα των οδηγών φορτηγών ε, όπου προτιμούν, προτιμούν ε, η αστυνομία να τους σταματήσει και να τους βάλει πρόστιμα γιατί οι εργοδότες τους, τους ε, πιέζουν πάρα πολύ να οδηγούν κουρασμένοι και να κινδυνεύουν να είναι κίνδυνος για το κοινό και τον εαυτό τους. Λοιπόν προτιμούν οι οδηγοί των φορτηγών στις διεθνείς μεταφορές, τις οδικές, να τους βάζουν πρόστιμα οι αστυνομικοί. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες θα πρέπει επίσης ε, ε, να καλλιεργήσουμε τον πολιτισμό της, ε, του σεβασμού και της υπακοής των κανόνων. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να σέβονται τους κανόνες οι οποίοι είναι σε ισχύ και να σέβονται γενικά τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Σε σχέση με το καμποτάζ είναι ένα ευαίσθητο θέμα φυσικά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό από το κοινό σαν κάτι το οποίο ε, δημιουργεί θέματα κοινωνικού dumping. Αυτό είναι αλήθεια παρά το γεγονός ότι μόνο του 2% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικά ανήκουν στην κατηγορία του καμποτάζ. Πρέπει όμως να αντιμεταπιστεί λόγω των κοινωνικών ανησυχιών, των κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως λόγω του ότι εάν το καμποτάζ είναι περιορισμένο ε, όταν παίρνουν κάποια εμπορεύματα εν πάση περιπτώσει στην επιστροφή τους μπορούν να κάνουν μόνο τρεις τάσεις σε επτά ημέρες και αυτός είναι ένας από τους λόγους ε, ε, για τους οποίους το ένα φορτηγό στα τέσσερα κινείται κενό στους αυτοκινητοδρόμους μας. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με συνολικό τρόπο και θα πρέπει να καταλήξει σε απλούς κανόνες οι οποίοι να είναι δίκαιοι και οι οποίοι να δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε τα του περιβάλλοντος με υπεύθυνο τρόπο και οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται σωστά κατανοητοί και φυσικά σεβαστοί. Μασιμιλιάνο Σαλίνη, σας ευχαριστώ. Κύριε Σεύκοβιτς, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε, λέει ο κύριος Σαλίνη, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τη διαχείρισή του στο σύστημα διαχείρισης, το ERTMS. Θα έπρεπε να είναι ενοποιητικός παράγων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα διευκόλυνε την διαλειτουργικότητα πέρα από τα σύνορα. Σε τεχνικό επίπεδο παραμένουν θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές του RTMS. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις γύρω από αυτό. Η πρώτη, θα συμφωνήσετε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στη σταθεροποίηση του ERTMS και των προδιαγραφών της. Και δεύτερον, θα διασφαλίσετε ότι η Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Υπηρεσία να είναι υπεύθυνη και για τις δύο πλευρές ε, αδειοδότησης και του υλικού και για το κινητό επίσης υλικό. Σας ευχαριστώ. Υπογραμμίσατε ένα θέμα σημαντικότατο για το μέλλον των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Το σύστημα ERTMS εκτιμάται από όλους τους εμπειρογνώμονες ότι είναι πολύ σύγχρονο ε, και τα σήματα κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα προχωρημένα τεχνικά και αυτή τη στιγμή σε εφαρμοστεί σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα τρένα ε, στα δίκτυα, περισσότερους επιβάτες, περισσότερα ε, εμπορεύματα και περισσότερη ασφάλεια. Βέβαια η ανάπτυξη του συστήματος αυτού ε, είναι κάτι το οποίο τώρα ολοκληρώνεται και θα θέλαμε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε γρηγορότερα από ό,τι προβλέπεται. Για να το πετύχουμε αυτό, η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να υπάρξει ένα σωστό διαχειριστικό σύστημα για την εφαρμογή του συστήματος και να πιέσουμε για την εφαρμογή του συστήματος αυτού στα κεντρικά σιδηροδρομικά ευρωπαϊκά δίκτυα, εκεί όπου χρειάζεται κυρίως περισσότερο ε, από ε, αλλού. Το σύστημα λοιπόν αυτό, αν ε, ίσχυε κάποια από τα τραχικά ατυχήματα που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο θα είχαν αποφευθεί, γιατί το σύστημα είναι καλύτερο και ασφαλέστερο. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι λοιπόν και για το κινούμενο υλικό, για τα βαγόνια δηλαδή και για το δίκτυο και για την σωστή εφαρμογή ε, του συστήματος ERTMS. Θα ήθελα επίσης να πάω ένα βήμα παραπέρα και να πω ότι θα έπρεπε ίσως να είναι ε, και υπεύθυνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των ανταλλακτικών των, ε, ε, των οχημάτων των συνδυοδρομικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε ότι έχετε εργαστεί σε μια απλή εργασία και όλοι χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ξέρετε τι θα πει να ζει κανείς με περιορισμένα ορισμένες αποδοχές. Ήμουνα οδηγό φορτηγού για 30 χρόνια και έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσα άδεια φορτηγά, υπήρχε περισσότερο καμποτάζ, αλλά με το νέο σύστημα κανόνων που ισχύει έχουμε ανοίξει τις πόρτες στους κακούς μέσα σε εισαγωγικά, αυτούς που φοράνε τα μαύρα καπέλα στα έργα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις ε, ε, πλαστές άδειες οδήγησης για τα φορτηγά. Από το ίντερνετ για 400 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει ένα διαβατήριο, ένα δίπλωμα οδήγηση επαγγελματικό και όλη την τεκμηρίωση. Μπορεί ένα άτομο να έχει τρία τέτοια διπλώματα και να οδηγεί 24 ώρες το 24 γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αστυνομία που να μπορεί να ελέγξει τη γνησιμότητα αυτών των αδειών Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται. Είναι ένας διεθνής κίνδυνος. Οι διαμεθοριακές μεταφορές είναι πολύ σημαντικές. Αλλά πλήττονται από αυτό το πρόβλημα. Ένας κανονικός ε, οδηγός θα πρέπει να καταγραφεί στην τοπική αστυνομία της περιοχής του. Αν όμως η εθνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ότι είναι πράγματι ε, νόμιμη και όχι πλαστή η άδειά του, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν ερώτημα αυτό, λέει ο κύριος Σεύκοβιτς. Ή μια δήλωση. Πιστεύω ότι δεν ήταν και η πρόθεσή σας γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά <clears throat> των οδηγών φορτηγών και εγώ δεν θεωρώ ότι οι οδηγοί οι οποίοι δεν κάνουν καμποτάζ είναι οι κακοί στο επάγγελμα αυτό. Κάνουν διεθνείς μεταφορές και γυρίζουν και πάλι στην βάση τους και προσπαθούν να βρουν κάποιο φορτίο στην επιστροφή ώστε να μην κυκλοφορεί το φορτηγό τους άδειο αν τώρα υπάρχουν καταχρήσεις του συστήματος. Συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Αλλά το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ το έχω τονίσει και πάλι είμαι έτοιμο να απλοποιήσω και να διευκρινίσω του κανόνε ώστε να υπάρχει σωστή εφαρμογή του. Αλλά η αστυνόμευση των κανόνων αυτών θα πρέπει να γίνει από τι εθνικέ αρχέ, γιατί αυτοί έχουν το δικαίωμα να το πράξουν. Και τωρα Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω για περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, ορεινές, παράκτιες, περιοχές που χρειάζονται δηλαδή επενδύσεις λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθήκων, αλλά και που έχουν ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Εγώ που την ε, Ουαλία, στην οποία δεν προβλέπονται διάδρομοι των Τσέντσι. Έχουμε ωστόσο ταυτόχρονα ανάγκη για καλές ε, διασυνδέσεις ε, σιδηροδρομικές. Είπατε ότι οι μεταφορές αφορούν τους πάντες. Ταυτόχρονα όμως μπορεί και να αποκλείουν κάποιους πολίτες. Πώς μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε ότι ε, επενδύσεις και υποστήριξη ορθές και σκόπιμες εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα για τις περιοχές με σεβασμό βέβαια και προς τον τουρισμό και τις περιοχές αυτές. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό όσο και δύσκολο, δυσεπίλητο ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι την ε, οπτική σας. Οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο ως παράγον συμπερίληψης, ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης οικονομίας, συμπερίληψης των, των ε, πόλεων στις περιφερειές τους σε εθνικό αλλά και διεθνές δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως, ε, εάν κοιτάξουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κυρίως δυστυχώς, δεν αρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ελήφθη μια απόφαση λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα και κυρίως σε σημεία συμφόρηση στους τομείς όπου προξενούνται σημαντικά προβλήματα με επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και τα σημεία όπου λείπουν οι σύνδεσμοι. Για την περίπτωση της Ουαλίας συγκεκριμένα που ρωτήσατε. Βεβαίως, εάν δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα των ε, διευρωπαϊκών δικτύων των μεταφορών θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση για την Ουαλία λόγω ακριβώς των κανόνων που έχουν υιοθετηθεί γιατί αυτοί ε, στοχεύουν ειδικά στην ε, αξιοποίηση κονδυλίων για τις προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ κύριε Σμαρτέζα. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, δεν απαντήσατε σε μία ερώτηση της κυρίας Ντέλη των Πρασίνων σχετικά με τη σύνδεση της γραμμής σιδηροδρομικής υψηλής ταχύτητας Λιών-Τορίνου. Είναι σκανδαλώδες να ξοδεύονται δημόσια χρήματα για τέτοιου είδους ε, ε, επενδύσεις είχε αποφασίσει έτσι και αλλιώς η Ιταλική κυβέρνηση να μειώσει κατά το 1 τρίτο τη συγχρηματοδότηση την εθνική. Ε, το κόστος από ό,τι φαίνεται όμως του έργου αυτού συνεχίζει να αυξάνεται. Η οικονομική κατάσταση στην Ιταλία και την Γαλλία σίγουρα δεν έχει βελτιωθεί και οι ανησυχίες για την αηφορία, την οικονομική και την ε, οικολογικοί ε, δυστυχώς αυξάνονται. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν εσείς το σύνολο του σχεδίου αυτού να το περάσετε από μια νέα οικονομική εξέλιξη, εξέταση συγγνώμη, ε, ή τουλάχιστον να δώσετε την ανάλυση αυτή σε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό και να μην δαπανίσετε περαιτέρω κοινοτικά χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς πολύ πιο απαραίτητους για την κοινοτικότητα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στην Ιταλία και στη Γαλλία, όπως επίσης και σε ε, ε, φόρα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω εδώ ότι ε, το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί. Ο κοινοτικός κανόνας λέει ότι πρέπει να σεβαστώ την απόφαση αυτή. Αυτό το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι σχετικά με την κατασκευή της υποδομής αυτής θα πρέπει να σεβαστούμε και άλλα, άλλες πλευρές και άλλα τμήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να υπάρξει σωστή διαβούλευση με το κοινό. Οι περιβαλλοντικοί κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Όλες δηλαδή οι πλευρές αυτές θα καταλήξουν στην ε, τελική έγκριση ενός τέτοιου ε, σχεδίου, ενός τέτοιου προγράμματος. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί λοιπόν όλοι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Τώρα, αν αρχίσουμε να τα συζητάμε όλα αυτά εκ νέου, φοβάμαι ότι θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και δεν θα μπορέσουμε να το κλείσουμε στη συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή της αποφάσεως αυτής σεβόμενη όλες τις πλευρές της κοινοτικής νομοθεσίας και σεβόμενη όλες τις ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει ακριβώς όπως είπα να γίνουν σεβαστές. Τελίτσκα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπατε κύριε υποψήφιε επίτροπε σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής use it or lose it. Αν δεν τα χρησιμοποιήσεις θα τα χάσεις. Ε, ήδη τέθηκαν ερωτήσεις για τα διόδια στην Γερμανία. Νομίζω ότι ε, το συζητάμε το θέμα αυτό εδώ και 25 χρόνια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και δεν το έχουμε πετύχει ακόμα αυτό. Και δεν έχω καταλάβει αν θα ξεκινήσετε εσείς την συζήτηση ε, για το κόστος αυτό το επιπλέον στις μεταφορές. Και όταν αναφέρεστε στον σεβασμό και ε, στην έλλειψη διακρίσεων, Ξέρουμε ότι οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται στην Γερμανία κατά κάποιο τρόπο ε, τεκμηριώνουν το επιπλέον αυτό κόστος. Ε, αλλά δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτό ε, να χρησιμοποιηθεί σαν αντιστάθμισμα για το κόστος των εσωτερικών μεταφορέων. Δεν έχω πρόβλημα με τα διόδια δηλαδή, με τα τέλη των διοδίων, αλλά η χρήση τους, σε πάση περιπτώσει, είναι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα γιατί όταν αυξάνει κανείς ε, ε, τις γραφειοκρατικές και τις οικονομικές επιβαρύνσεις ταυτόχρονα θα παίρνει και μέτρα ελάφρυνσής τους. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Και είμαι σίγουρο. ότι μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας για μια πολύ αυστηρή επαλήθευση της στήρησης του κανόνα use it or lose it, αξιοποίησε ή χάνει την ευκαιρία σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί γιατί είναι πολύ περιορισμένοι δημοσιονομικοί πόροι. Και το, η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντικά, έχουμε, σημαντική, έχουμε πάρα πολλά μεγάλα έργα και θα πρέπει να αποδείξουμε και να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα αξιοποιούν τους πόρους εγκαίρως ή θα κινδυνεύουν να τους χάσουν. Και βεβαίως εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί για δε την κατάσταση τη σχετική με τα διόδια στη Γερμανία. Όπως είπα, αφενός μεν χαίρομαι που ξεκινάει, που ανοίγει η συζήτηση στη Γερμανία. Ο, η αναζήτηση δηλαδή της ε, εσωτερήκευσης εξωτερικού κόστους, γιατί η Γερμανία έχει την τεράστια υποδομή ως χώρα. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και να κλείνουν γέφυρες και να μην υπάρχει σωστή συντήρηση ορισμένων αυτοκινητοδρόμων. Χαίρομαι λοιπόν που η συζήτηση αυτή άρχισε συζήτηση η οποία αφορά και το πώς μπορεί να εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστος της ε, χρήσης των ε, οδικών υποδομών. Όπως είπα, έχει τεράστια σημασία για μένα η αρχή ο πληρώνει και η αρχή της απαγορεύσεων διακρίσεων. Αυτό θα είναι σαφέστατο εκ μέρου μου, θα καθίσετε σαφέστατο όταν βλέπω, όταν δω συγκεκριμένα το διατακτικό του νόμου που πρόκειται να καταθέσει η γερμανική κυβέρνηση, θα το εξετάσω με απόλυτη αυστηρότητα. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεύκοβιτς, για τις ε, απαντήσεις Θα ήθελα να επισημάνω ότι με χαρά λαμβάνω το λόγο μετά τον συνάδελφο ο οποίος είχε ε, το συντονισμό του προγράμματος για τη Βαλτική. Θα περιμένετε, φαντάζομαι, θα αναμένετε αρκετή υποστήριξη από την Επιτροπή μας ε, για το θέμα της Βαλτικής. Εμείς έχουμε μια ισχυρή βρετανική στηρητική ε, ομάδα στην ε, ομάδα των στηρητικών μεταρρυθμιστών που όμως αποσιάζει αυτή τη στιγμή ο εκπροσωπός της διότι βρίσκεται σε μια ε, διάσκεψη στην Βρετανία σε ένα συνέδριο, αλλά έχω αναλάβει εγώ να τον εκπροσωπήσω. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για την πρωτοβουλία για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες που μπορεί να παρεμποδιστεί από διάφορα μέτρα ε, που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν λοιπόν να επιταχυνθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είχατε και την πιο εύκολη ερώτηση εγώ να υποβάλω. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι και σας ευχαριστώ θερμά. Για την ερώτηση λοιπόν αυτή. όποιος θέλει να προωθήσει ένα αίσιο μέλλον, ένα καλό, μια καλή προοπτική για τους ευρωπαϊκούς εθέρες, θα πρέπει να αισθάνεται μια κάποια δυσφορία για το ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με τα λεγόμενα FABS, την ε, εξασφάλιση εννέα εδαφικών στοιχείων, που χωρίς να είναι ιδεώδης λύση γεννούν νέες και ποικίλε ευκαιρίες για πιο σύντομους δρόμους, για πιο, σύντομες δρομές δηλαδή για εξοικονόμηση χρόνου, πόρων, εκπομπών στις αεροπορικές πτήσεις. Όπως είπα, αυτό ισοδυναμεί σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος. Όπως είπα, Μέχρι τώρα η πρόοδος είναι μάλλον περιορισμένη και αισθανόμαστε μια κάποια απογοήτευση. Θα προτείνω λοιπόν καταρχάς να αξιοποιηθούν περισσότερο τα κριτήρια αποτελεσματικότητας ή απόδοσης καλύτερα, όπου θα πρότεινα στα FAPS να ε, προσμετράτε ε, το κριτήριο της απόδοσης και πόσο θα μπορούσε ακόμη να συντομεύσει μια πτήση, να περιοριστούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πτήσης μέσα σε ένα ΦΑΠ που θα είναι συγκρίσιμο με το ΦΑΠ κάποιου άλλου και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα υγιή ανταγωνισμό που θα δείχνει πώς ένα ΦΑΠ έχει καλύτερα αποτελέσματα από κάποιο άλλο και πόσα χρήματα χάνονται κάπου αλλού. Και βεβαίως Εάν δούμε ότι ε, υπάρχει μια συνεχιζόμενη ε, ε, παραγνώριση των αρχών των ΦΑΠΣ, τότε θα πρέπει να διδαρχήσουν και διαδικασίες επί Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουιέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτς, είμαι εδώ αμέσως μπροστά σας. Ως ε, ο τελευταίος ομιλητής από τους σοσιαλιστές και αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα ήθελα να σας τονίσω ότι μετά από σχεδόν τρεις ώρες, μια μαραθώνια ακρόαση, ξέραμε ότι ήσασταν εξαιρετικός διπλωμάτης, το είδαμε από το βιογραφικό σας, αλλά είσαστε και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για τα θέματα μεταφορών και δείχνετε σημαντικό ενθουσιασμό για τα θέματα αυτά. Είδα την ε, γραπτή σας απάντηση και είχα κάποια ερωτήματα, αλλά τα έχετε απαντήσει όλα. Μπορείτε λοιπόν να χαλαρώσετε, ας αφήσουμε τις μεταφορές και πέστε μου το εξής. Τα επόμενα χρόνια, ως ένας γείτονας από την Κεντροανατολική Ευρώπη με την ιστορία της χώρας σας, πώς, θα είναι, πώς θα είναι το μέλλον της ε, Ευρώπης σε επίπεδο μεταφορών. Τι μπορούμε να κάνουμε που είναι το πιο σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ λέει και ο κύριος Σεύκοβιτς για την πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό, είμαι αισιόδοξο από αυτή την άποψη. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν πολύ δύσκολη εποχή βρεθήκαμε στο χείλος της κατάρρευσης ουσιαστικά της διαδικασίας ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Αλλά όταν συζητάμε για το πού βρισκόμασταν πριν από 25 χρόνια πριν και πού βρισκόμαστε τώρα, είναι η ιστορική πρόοδος που έχουμε επιτύχει και παρά τα τελευταία χρόνια της κρίσης δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο έχει αλλάξει η Ευρώπη και πόσο έχουμε προχωρήσει και πόσο πολύ πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά τα θέματα αυτά. Εγώ μεγάλωσα στην Πρατισλάβα πίσω από το συνδρόμο παραπέτασμα. Νόμιζα όταν ήμουν νέο ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να φτάσω στην Αυστρία, θα με σταματούσαν στα σύνορα. Είναι ένα θαύμα αυτό που έχει συμβεί και πρέπει να το ομολογήσω. Το καταπληκτικό είναι ότι τα παιδιά μας το παίρνουν για δεδομένο. <clears throat> Θεωρούν δεδομένο ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν υπάρχουν εκεί έλεγχοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει. Πρέπει και εμείς για τις μεταφορές να κάνουμε το ίδιο. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή σας είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη και προσφελωμένη να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή αυτή που έχουν περάσει όλη τους την καριέρα στον τομέα των μεταφορών. Έχω συναντήσει πολλούς από εσά και ξέρω πόσο υποστηρίζετε την Ευρώπη και πόσο θέλετε να εργαστείτε για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά ένα ε, ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο χωρίς σύνορα, χωρίς ελέγχους, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προστατευτισμό, μία μονάχα ενιαία Ευρώπη μεταφορών. Υπάρχει όμω και μια ακόμα ερώτηση παρά τα χειροκροτήματα. Η κυρία Λουκατσιεύσκα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάω κατευθείαν στην ερώτησή μου και ότι ο υποψήφιος επίτροπος έχει απαντήσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Θα τη θέσω. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση τώρα για το καμποτάζ ε, όπως αυτή επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα πρέπει να πράξουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τις οδικές μεταφορές, να ε, ενισχύσουμε το δυναμικό τους την παραγωγικότητά τους και τι πρέπει να κάνουμε για να ε, εφαρμοστούν επιτέλους οι διατάξεις οι οποίες δεν βρίσκονται ακόμη ενισχύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τους ε, οδικούς μεταφορείς ε, που δεν έχουν ακόμα μπορέσει να λύσουν το πρόβλημα της διαμετακόμισης λόγω του εμπάργου που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της διαμετακόμισης είναι προφανώς πολύ ε, λεπτό, έχει πολλές ε, συνέπειες και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς πολύ μεγάλο τμήμα των μεταφορών μας περνάει μέσα από αυτό. Πρέπει να απλουστεύσουμε και να διευκρινίσουμε τους κανόνες νομίζω, διότι Πρέπει πάνω απ' όλα να αποκαταστήσουμε το αίσθημα της κοινωνικής ασφάλειας για τον οδηγό του φορτηγού. Πρέπει και είναι πολύ σημαντικό και εδώ θα πρέπει να κληθούν και οι εθνικές αρχές να ενισχυθεί η επιβολή, η εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν. Η τεχνολογία επίσης, η παραδείγματι, στο, στις μετρήσεις. Ο υπολογισμός ε, του εάν τηρούνται οι κανόνες, ο ψηφιακός ταχογράφος ή οι νέες τεχνολογίες οι οποίες και χάρη νέο σύστημα, στα νέα συστήματα πλοήγησης και το δυναμικό που προσφέρουν οι δορυφόροι ε, στην Ευρώπη μπορεί να είναι ένα ζήτημα αξιολόγησης. Και όταν η Ευρώπη έχει το, την πρώτη θέση, την πρωτορική θέση στην επιμελητία, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν καλύτερα το ε, χρόνο οδήγηση στην διαχείριση του φορτίου, την επιμελετειακή ολοκλήρωση σε ένα διατροπικό είδος μεταφορών, σε ένα χώρο μεταφορών που οικοδομούμε στην Ευρώπη. Όπω είπα, ένα στα τέσσερα φορτηγά κυκλοφορεί κενό φορτίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσουμε. Για δε τα προϊόντα που εξάγονται προ τη Ρωσία είναι απαράδεκτη κατάσταση που έχει επέλθει με το εμπάργκο. Στο προσεχές, ε, στην προσεχή συνεδρία τη Επιτροπή θα το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Θα βρούμε μια λύση συνεργασία με τι ρωσικέ αρχέ, γιατί δεν είναι δυνατό να υποφέρουν οι οδηγοί των φορτηγών μας επειδή υπάρχουν εντάσεις στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, απαντήσατε σε 38 απαντήσεις. Έχετε ακόμα 5 λεπτά για να πείτε τα τελευταία και καταληκτικά λόγια. Thank you Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, uh, Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι από αυτό που ακούστηκε επιβεβαιώθηκε ότι και η Επιτροπή Μεταφορών και η Επιτροπή Ήτρε είναι ιδιαίτερα ισχυρές στην αφοσίωσή τους ε, για την Ευρώπη στην Ευρώπη και στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί από εσά έχετε εργαστεί στα θέματα των μεταφορών εδώ και αρκετό καιρό. Είσαστε αρκετοί που ήσασταν υπουργοί μεταφορών, κάποιοι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικοί στις μεταφορές εδώ και πολλά χρόνια. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί στον τομέα των μεταφορών τα επόμενα χρόνια, η επόμενη φάση χρονική θα είναι ιδιαίτερος κρίσιμη. Εδώ μπορώ να το συνδέσω αυτό με τις ερωτήσεις τις οποίες ε, μου θέσατε και εσείς. And uh, the future of uh, transport area. Νομίζω ότι εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ε, αυτό που πιστεύω για τον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πέντε χρόνια. Απλά κριτήρια. Καταφέρατε ε, να ανακάμψετε, καταφέρατε να δημιουργήσετε νέες θέσεις απασχόλησης, καταφέρατε να προπαρασκευάσετε την Ευρώπη στην παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποιημένη οικονομία, να την κάνετε πιο ανταγωνιστική. Το κάνατε αυτό με τον ευρωπαϊκό τρόπο, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον. Αηφόρος ανάπτυξη με υψηλά κοινωνικά κριτήρια. Φυσικά αυτές οι ερωτήσεις που θα τεθούν μετά από πέντε χρόνια δεν θα είναι εύκολες ερωτήσεις γιατί κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα είναι κριτής Πάντως πιστεύω ότι έχουμε τα μέσα για να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω με τις κοινέ μας προσπάθειες θα το καταφέρουμε. Ξέρετε πολλοί από εσά που έχουμε συνεργαστεί στην προηγούμενη περίοδο ότι είμαι υπέρμαχος της σωστής σχέσεις και συντονισμού ανάμεσα στα δύο αυτά κοινοτικά όργανα. Εγώ είχα συνεργαστεί ε, με την διάσκεψη των προέδρων των, ε, προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τους προέδρους της επιτροπής σας δηλαδή και νομίζω ότι θα συνεχίσω προς την κατεύθυνση αυτή μια σωστά ε, διαρθρωμένη στενή συνεργασία. Μένει πάρα πολλά να γίνουν η ατζέντα που έχουμε μπροστά μας, ε, η κοινή είναι τεράστια. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι κεράστια. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε ε, ε, να το κάνουμε από κοινό και αν με στηρίξετε θα εκμεταλλευτώ τη στήριξή σας αυτή αλλά σε συνεργασία μαζί σας πάντα. Ja, mit diesem statement... Και με αυτή τη δήλωση έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ακρόασης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους τους βουλευτές, για τις εμπεριστατωμένες σας ερωτήσεις. Έχουμε καλύψει ένα ευρύ πεδίο της πολιτικής μεταφορών και διαστήματος. Ευχαριστώ και τον υποψήφιο επίτροπο, τον Μάρο Σεύκοβιτς, για τις απαντήσεις που μας έδωσε και για τις θέσεις που πήρε. Υπενθυμίζω στους συντονιστές και τους αντιπρόεδρους της ε, επιτροπή μας ότι η συνεδρίαση για την αξιολόγηση της ακρόασης θα γίνει στο Α1G2 στις 9.30 και θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και τους ε, διερμηνείς για τη θαυμάσια εργασία τους και την εγκαρτέρησή τους και τους ευχαριστώ γιατί ξεπεράσαμε λιγάκι και το χρόνο που προβλεπόταν για την ακρόαση. Βλέπετε ότι έχει πράγματι εκτιμηθεί το έργο σας και σας εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ. Γεια σας.